Bueno, buenos días. Vamos a ir empezando porque si no... Καλή σας μέρα. Ας ξεκινήσουμε. Γιατί αλλιώς θα περάσει η ώρα και μετά άντε να τελειώσει. Ξεκινάμε μια ακόμα μέρα με πολύ ενθουσιασμό. Σημείο 12 της Μέσιας Διάταξης, γνώσεις για τη θάλασσα 2020, βελτίωση της χαρτογράφης του βυθού για αλευτικού σκοπούς. Θα θυμάστε ότι η Κομισιόν έχει, είχε υποβάλει μια πράσινη βίβλο για τη γνώση του θαλάσσιου ε, βυθού και εμεί αποφασίσαμε και ορίσαμε ως εισηγήτρια την κυρία Πατράου ε, να εκδώσουμε μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για να δούμε πώς μπορούμε μέσω αυτού του προγράμματος να προωθήσουμε τη βιώσιμη αλία. Ε, η κυρία Πατράου θα μας παρουσιάσει την έκθεση. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. Και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Επιτροπής. Γιατί σχετίζεται με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πράσινη βίβλο της ε, Κομισιόν για τη γνώση του θαλάσσιου βυθού του 2020. Ε, πρόκειται για μια πράσινη βίβλο πολύ ολιστική, πολύ πλήρη, σφαιρική. Ε, μέσα σε αυτήν η Αλία έχει αντιπροσωπεύει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι, σχεδόν μηδενικό. Το έγγραφο αυτό όμως ε, αποτελεί πυλώνα της ε, γαλάζιας οικονομίας ε, προς την οποία έχει προσιλωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάσσεται πολύ εύκολα στους στόχους στρατηγικής 2020, οπότε είναι σημαντικό και η Αλία να βρει τη θέση της μέσα στις κατευθυντήρες δαμές προς προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι η Αλία δέχεται επίθεση από διάφορα μέτωπα και με διάφορους τρόπους. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό να δείξουμε ποια είναι η θέση της Αλίας σε ένα τέτοιο έγγραφο όπως η Πράσινη Βίβλος Κομισιόν. Ο στόχο τη Κομισιόν με την Πράσινη Βίβλο είναι να δημιουργηθεί ένας ε, χάρτης ε, συνεχούς πολλαπλής ανάλυσης, ψηφιακός χάρτης του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων ω το 2020. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και πολύ επιστημονικό έργο ευρεία κλίμακας, το οποίο αποσκοπεί να διασφαλίσει τη διάθεση πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα ε, ενδιαφερόμενων φορέων, ε, στοιχεία τα οποία θα αποκτηθούν, θα συλλεχθούν, θα διασυνδεθούν και θα ε, τεθούν στη διάθεση του κοινού με διάφορους τρόπους θα σας εξηγήσω σε λίγο. Η Αλία πρέπει λοιπόν να εκφράσει την άποψή της Ε, εξηγώντα πώς μπορεί να συνεισφέρει στην ε, υλοποίηση του σχεδίου και πώς μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το σχέδιο. Όπως είπα και σε προηγούμενες παρουσιάσεις, εδώ στην Επιτροπή έχω διαρθρώσει ε, το, την έκθεσή μου σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Πρώτον, ε, τύποι δεδομένων και πηγές δεδομένων. Δεύτερον, απόκτηση και διαθεσιμότητα δεδομένων. Τρίτον, ε, αποτελεσματική συλλογή και διασύνδεση των δεδομένων και τέταρτον ε, πώς μπορούμε να αποφεληθούμε από την επεξεργασία και την ερμηνεία των δεδομένων. Με βάση αυτή τη ε, δομή συνέταξα και την έκθεσή μου. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, πηγές ε, πληροφοριών και τύποι δεδομένων. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που κατέχουν δεδομένα σχετιζόμενα με την αλία και θα μπορούσαν να, όλα αυτά τα δεδομένα να ενταχθούν στη χαρτογράφηση. Ορισμένοι από αυτά τα δεδομένα έχουν ήδη συλλεγεί και έχουν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του πίνακα για τη συλλογή δεδομένων ε, αλίας κυρίως. Υπάρχουν όμως και άλλες πηγές οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, τα συστήματα παρακολούθησης της αλληλευτικής προσπάθειας, πολύ χρήσιμα αυτά τα δεδομένα, ε, δεδομένα από τα ηλεκτρονικά ημερολόγια καταστρώματος, ε, αρχεία ε, των παρατηρητών αλίας στα σκάφη κλπ. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για την αλία και αποκτώνται στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνών ε, και προγραμμάτων. Δεύτερο σημείο, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την απόκτηση και διαθεσιμότητα των δεδομένων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί για την διευκόλυνση αυτής της ε, διαθεσιμότητας, να καθοριστούν όροι και επίπεδα πρόσβασης διαφορετικά για κάθε τύπο στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης τη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και εδώ μην αγνοήσουμε και τα εμπορικά συμφέροντα τα οποία σχετίζονται με την αλία. Δεδομένου ότι η απόκτηση, η συλλογή μάλλον των δεδομένων, η διαχείριση των πληροφοριών έχουν προκύψει από επιστημονικά προγράμματα πολύ συχνά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει αυτή την συλλογή και, και διαθεσιμότητα οπότε ε, λογικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να τα καταστήσει δημόσια. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που έχουν αποκτηθεί με ιδιωτική χρηματοδότηση, εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια άλλη μεθοδολογία, θα πρέπει να ζητείτε η άδεια ε, αυτών των φορέων που τα έχουν χρηματοδοτήσει, που έχουν τη συλλογή τους, προκειμένου να γίνουν, καταστούν δημόσια. Όταν τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τα έσοδα των συλλεκτών, αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια ε, ως ε, προϊόντα δεδομένων και όχι ως ε, δέντρο δεδομένα αυτά καθεαυτά. Ε, Πρέπει επίσης να γίνεται υποχρεωτικά αναφορά στην πηγή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με τον συλλέκτη των δεδομένων και να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες ή ακόμα και τα ε, μη επεξεργασμένα δεδομένα. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων για, για το στόλο ε, θα πρέπει να γίνεται με προστασία της, ε, του απόρριτου. Για παράδειγμα, ε, τα ημερολόγια αλίας, ε, οι εκθέσεις των παρατηρητών και τα στοιχεία του VMS θα πρέπει να αποφύγουμε να δίδουν στοιχεία για συγκεκριμένα πλοία, για παράδειγμα το όνομα ή τον αριθμό καταχώρησης του πλοίου. Το εμπορικό απόρριτο και εμπιστευτικότητα μπορούν να ενισχυθούν μέσω της ε, χρήσης ε, ε, ομαδοποιημένων δεδομένων. Με αναφορά στον τύπο αλληλείας, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και βέβαια με χρονική διαφορά ανάμεσα στη συλλογή και τη δημοσιοποίηση διαθεσιμότητα των ε, των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο χρόνος. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια χρονική απόσταση ανάμεσα στη συλλογή τους και την ε, θέση σε διαθεσιμότητα, την δημοσιοποίησή τους. Τώρα, τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλογεί από κρατικούς φορείς των κρατών μελών, για αυτά θα πρέπει να φύσταται ένα σε αριθμός όρων σε ό,τι αφορά το πώς θα γίνονται, ε, πώς θα γίνει η δημοσιοποίησή τους. Δηλαδή θα πρέπει να ακολουθούν το ίδιο φορμάτ έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να δημοσιοποιούν συγκρίσιμα στοιχεία. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε κοινού όρους σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ε, υποχρεωτικές ε, παραμέτρους, ελάχιστες παραμέτρους για τον ε, τρόπο της παρουσίασης των δεδομένων. Για στοιχεία τα οποία έχουν συλλεγεί από επιστημονικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, και κατά 50% τουλάχιστον συγγνώμη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένους τρόπους. Στο πλαίσιο των επιστημονικών προγραμμάτων είναι λογικό να δίδεται ε, ένα εύλογο χρονικό διάστημα στους ε, επιστήμονες ε, προκειμένου να ε, δημοσιεύσουν τις εργασίες τους πριν τα στοιχεία αυτά γίνουν δημόσια. Λογικό είναι και πρέπει να γίνει σεβαστό το επιστημονικό έργο. Ε, πρώτα θα πρέπει να δημοσιεύονται τα πορίσματα της έρευνα και μετά τα ίδια τα στοιχεία. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και την ερμηνεία των δεδομένων. Αυτή περνάει από τον ε, έλεγχο της ποιότητας ε, των δεδομένων καταρχήν. Πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο έτσι ώστε να μπορέσουν να διορθωθούν σωστά τα δεδομένα που έρχονται από διάφορα κράτη-μέλη. Ε, είναι απαραίτητο λοιπόν να ακολουθούνται πρωτόκολλα, κοινά μοντέλα, ενοποιημένα μοντέλα για την ε, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ένα φορμά τρόπος παρουσίασης, κοινός τρόπος παρουσίασης των δεδομένων. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο για τη συλλογή δεδομένων τομέα τη αλίας, το οποίο, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη. Ο τρόπο με τον οποίο θα διατίθενται τα δεδομένα θα εξαρτάται από την πολυπλοκότητα αυτών. Ορισμένε απλέ παράμετροι θα μπορούσαν να δίδονται για, με δεδομένα μη επεξεργασμένα, ενώ κάποια πιο συγκεκριμένα και πιο ειδικά στοιχεία θα χρειάζεται, κάποιες πιο ειδικέ παράμετροι θα πρέπει να παρουσιάζονται με βάση στοιχεία επεξεργασμένα ε, ή προϊόντα δεδομένων. Διάρθρωση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση ε, της ποιότητας, της ποσότητας και της ε, τρόπου των δεδομένων. Και με, έτσι ώστε μετά να μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αξιολογεί τακτικά και αυτή τη διαδικασία. Τελευταίο σημείο σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των δεδομένων. Ε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την σημασία της διακυβέρνησης και της λειτουργίας. της διαδικασίας το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Παρατήρησης ε, Δεδομένων ΕΜΟΤΝΕ θα πρέπει να ε, ηγηθεί της προσπάθειας, πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πρόσθετη θεματική ομάδα για την αλία μέσα στο M.O.D.Net η αλία στην ομάδα που πρόσφατα δημιουργήθηκε για τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εγώ πιστεύω η πρώτη είναι η καλύτερη λύση. Δικαιολογείται η δημιουργία μιας ειδική θεματικής ομάδας για την αλία. Πέραν αυτού, είναι σημαντικό αυτή η πλατφόρμα του M.O.D.Net να συνδεθεί με την θαλάσσια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης της Γης ε, για να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των δεδομένων και να συνδέονται τα δεδομένα μεταξύ τους, δηλαδή ε, τα δεδομένα της παρατήρησης από δορυφόρο με τα δεδομένα της αλίας. Δεν θέλουμε αλληλεπικαλύψεις, δεν μπορούμε να αυξήσουμε το κόστος, πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τους πόρους που ήδη διαθέτουμε. Να επενδύσουμε σε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση αυτών που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Αποφεύγοντας αλληλεπικαλύψεις και πρόσθετο κόστος. Να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους. Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία θα πρέπει να ενισχυθεί και με πληροφορίες σχετικές με την αλληλεία μέσω μιας ενός προγράμματος δράσης που θα έχει συγκεκριμένους στόχους μακροπρόθεσμους και ε, μεσοπρόθεσμους. Δεν αρκεί να έχουμε σχέδια στα χαρτιά, δεν αρκούν οι προθέσεις, οι καλές προθέσεις, χρειαζόμαστε πρόγραμμα δράσης. Το πρόγραμμα δράσης αυτό θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο, με στόχους που θα έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων και με αξιολόγηση, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν. Γιατί αλλιώς τα μεγάλα σχέδια και τα μεγάλα λόγια θα μείνουν στα χαρτιά. Χρειάζεται βέβαια και ε, επαρκή σηματοδότηση αυτό το πρόγραμμα και εγγύηση συνέχειας, μακροπρόθεσμα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε πολιτικές βραχυπρόθεσμες με πολύ στενό ορίζοντα Χρειάζεται ένα, μια χρηματοδότηση μέχρι το 2020 έτσι ώστε πραγματικά να καταλήξουμε σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι ε, αποδοτικά για την βιώσιμη εκμετάλλευση του βυθού και ιδιαίτερως της αλίας. Συγγνώμη, της θάλασσας και ιδιαίτερως της αλίας. Χρειάζεται λοιπόν χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του project το 2020. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές της έκθεσής μου. Σας είχα ήδη παρουσιάσει ένα προσχέδιο. Είχαμε ανταλλάξει απόψεις καταρχήν και μετά σας είχα ε, υποβάλει το προσχέδιο της ε, έκθεσης που είχα προετοιμάσει. Ε, νομίζω ότι με είχατε ήδη στηρίξει. Προφανώς ε, έχω εντάξει ήδη ε, τις πρώτες σας παρατηρήσεις στο κείμενο. Είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω κάποια πρόσθετα σχόλια. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Μέσνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτριά μας. Πρέπει να πω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή, διεξοδική. Ασχοληθήκαμε με το θέμα στην Επιτροπή Αλίας σε μια ακρόαση οργανωμένη πολύ καλά από εσά και πράγματι χρειαζόμαστε πιο πολλές γνώσεις και δεδομένα για την αλία και τη χαρτογράφηση του βυθού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό προϋπόθεση για να προχωρήσουμε, γιατί μιλάμε για τη γαλάζια ανάπτυξη και σε αυτά τα πλαίσια η αλία έχει μεγάλο μερίδιο. Για να προχωρήσουμε περισσότερο θέλουμε καλύτερα δεδομένα, καλύτερες πληροφορίες, γενικότερα και πρέπει όχι μόνο να ζούμε, αλλά και να αξιοποιήσουμε περισσότερο τους ωκεανούς. Γι' αυτό προϋποτίθενται περισσότερα δεδομένα, αλλιώς δεν γίνεται. Εμένα μ' αρέσει αυτό γιατί είμαι πολύ υπέρ της ολοκληρωμένης πολιτικής αλίας και είναι η αλληλεία ένα, μια άμεση δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και γι' αυτό το αναφέρεται και σε μια αιτιολογική σκέψη και μου άρεσε πολύ. Είναι πολύ παλιά δραστηριότητα αυτή. Η ανταλλαγή δεδομένων είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε ε, επιστημονική προσέγγιση. Υπάρχουν πολλά δεδομένα, αλλά δεν είναι τυποποιημένα όλα, ούτε υπάρχει ανταλλαγή τους. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και πολύ σωστά το αναφέρει η συγκήτρια. Έχουμε την πλατφόρμα του MOVNet και πρέπει αυτή να βελτιωθεί, αλλά πρέπει να παίρνουν και δεδομένα με τη σωστή μορφή. Χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο την έρευνα και αυτό το λέτε για να αποκτήσουμε περισσότερα δεδομένα και πάνω απ' όλα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε καλά τα δεδομένα και να γίνεται σωστή ε, επεξεργασία τους. Ε, οι ωκεανοί μόνο σε μικρό ποσοστό έχουν εξερευνηθεί. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό ε, ωκεάνιο και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Έχουμε δεδομένα, στο μέλλον θα έχουμε και περισσότερα το αναφέρει αυτό η συγγήτρια, είναι σε δημόσια ιδρύματα, σε ιδιωτικά, εν μέρη βρίσκονται και στα χέρια των επιχειρήσεων, αλλά ακόμη δεν είναι εύκολη η ε, στοχευμένη και ε, συντονισμένη ανάκλησή τους. Είναι λοιπόν σωστό να μπορούμε να τα παίρνουμε και για να τα παίρνουμε θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο για να τα διαβιβάσουμε περισσότερο. Ε, κάποιος που ερευνά μια επιχείρηση που έχει ε, δεδομένα μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζει και άλλα δεδομένα ή να έχει και κοινέ βάσεις δεδομένων για να, να γίνεται ε, η ανάκληση από όλους. Και αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε και σωστά το λέει η συγγήτρια. Είναι απόλυτα λογικό να πούμε ότι την ε, πρόθεση της έρευνας και της συλλογή δεδομένων τη συνδέομαι με την ανάγκη και την προϋπόθεση να διαβιβάζονται τα δεδομένα παραπέρα, ιδιαίτερα στον τομέα της αλίας, για να χρησιμεύουν καλά. Και θα πρέπει και να το τυποποιούνται, να εναρμονίζονται τα δεδομένα αυτά για να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις και τη διπλή δουλειά. Και αυτό το λέει η γι' αυτό σας είπα ότι η έκθεσή της είναι εξαιρετική. Ε, η ανάκληση να γίνεται σωστά. Γενικά η αλληλεία και τα δεδομένα της αποτελούν σημαντικό κομμάτι της γαλάζιας ανάπτυξης. Η χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας είναι σημαντικό. Η Κομισιόν εδώ και καιρό είπε ότι χρειάζεται για να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό για να εξερευνήσουμε καλύτερα τους ωκεανούς. Τα δεδομένα είναι το νόμισμα του μέλλοντος θα μπορούσαμε να πούμε για τη γαλάζια ανάπτυξη ως ένα βαθμό. Γι' αυτό όλα αυτά τα υποστηρίζω γιατί η εισηγήτρια ζήτησε υποστήριξη και μπορώ να τη διαβεβαιώσω ότι έχει την υποστήριξη των φιλελευθέρων. Ενδεχομένως ε, θα κατατεθούν κάποιες μικροτροπολογίες συμπληρωματικές, όχι για να αλλάξουμε την ουσία της έκθεσης. Ευχαριστώ. Συνεργαζόμεθα πολύ καλά και με τη θαλάσσια ε, χωροταξία. Συχνά δηλαδή θα ασχοληθούμε και θα συνεργαστούμε μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Κρίστιανσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Αρσένη, του Σκιώδους από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, είναι, έχει δύο φακέλους σε άλλη επιτροπή όπου και εκεί είναι σκιώδης έτσι στην ΕΝΒΗ. Λοιπόν, θα παρουσιάσω εγώ αυτά που θα πει. Χαιρετίζω την έκθεση της εισηγήτριας, τη συγχαίρω για τη σκληρή δουλειά που έκανε. Υπάρχουν πολλά σημεία συμφωνίας αλλά και διαφωνίας με την έκθεση της εισηγήτριας. Χαιρετίζω την ένταξη των πολλών Εβραίων δεδομένων για την αλληλευτική δραστηριότητα στην Ένωση ε, σε έναν χάρτη ψηφιακό για το βυθό των θαλασσών. Ε, είναι πολύ σημαντική πηγή που θα χρησιμοποιείται από την ISIS όταν θα γνωμοδοτούν για θέματα διαχείρισης ελίας. Ε, όταν χαρτογραφούμε τις ελιευτικές δραστηριότητες, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό υπογραμμίζω ότι το GPS, VMS και τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται και στη βιομηχανική αλία και στην αλία μικρής κλίμακας. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να τυποποιούνται, να επαληθεύονται και να ελέγχονται. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών στον τρόπο συλλογής των δεδομένων την επεξεργασία τους, τη σύνταξή τους και η διαδικασία συλλογής ε, και όπως και οι πρωτοβουλίες εξαρτώνται από τη συνέχεια και την προβλεψιμότητα κατάλληλης χρηματοδότησης μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Διαφωνώ όμως ε, στο θέμα της ε, προστασίας του απορρίτου των δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται και χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να διατίθενται δημόσια ή τέλος πάντων θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση στην πρόσβαση. Ε, πρόκειται για δημόσια αγαθά, ε, εδώ και ιδιαίτερα αυτό είναι σημαντικό σε περίοδους κρίσης όπου χρησιμοποιούνται χρήματα των φορολογουμένων για τη συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα που προκύπτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσια ε, και η χρήση εμπορικών ε, απορρίτων είναι κάτι το απαράδεκτο. Αυτό που είναι εμπορικό συμφέρον για τον Αλιέα είναι ένα ε, στοιχείο ε, εμπιστευτικό, αν θεωρούνται και τα ετήσια ελιεύματα εμπιστευτικά. Ε, ποιος θα ωφεληθεί από μια δημόσια πηγή ε, ποιοι ορισμοί θα υπάρξουν. Οι παράγραφοι 7, 9, 11, 12 είναι ιδιαίτερα προβληματικές και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει πάντοτε να συμμορφούνται με την Σύμβαση του Άρχους για την πρόσβαση στην πληροφορία, τη δημόσια συμμετοχή τη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα της 15ης Ιουνίου του 2008. Τέλος, να υπογραμμίσω ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, οικοσυστήματα, θαλάσσια, ε, ε, χώρους αναπαραγωγής των αποθεμάτων που θα πρέπει να προστατεύονται μέσα από ε, την θέσπιση περιοχών θαλάσσιων προστατευόμενων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω την εισηγήτρια το εξής η Βρετανική κυβέρνηση θα υποχρεούται να δίνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την το θαλάσσιο βυθό στα χωρικά υδατά της και θα υπάρξει διαδικασία επιπαραβάση αν δεν το κάνουμε, θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη χθεσινή ψηφοφορία, όπου ψηφίσαμε για να ε, επιδοτήσουμε τις ε, τράτες ε, και λαμβάνοντας το αποτέλεσμα στα αποθέματα. Δεν θα ήταν καλύτερα να ε, ε, ε, επιδοτήσω τα λιευτικά σκάφη για να πηγαίνουν και να λιεύουν τα δεδομένα παρά τα ψάρια, ούτως ώστε ο πλοίαρχο να κάνει μια έρευνα για συγκεκριμένη περιοχή του βυθού της θάλασσας και να πληρώνεται γι' αυτό. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Ευχαριστώ κυρία Λιβάνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια Πρόκειται όντως για ένα σημαντικότατο θέμα. Βέβαια τα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν ενδιαφέρονται για τα σύνορα των κρατών μελών, οπότε αυτό αν θέλετε είναι η πρώτη παραδοχή μας όταν μιλάμε για το βυθό της θάλασσας και τους ωκεανούς. Έχει νόημα λοιπόν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν εδώ και αν θέλουμε να προστατεύσουμε κάποια ευάλωτα οικοσυστήματα, πρέπει να έχουμε δεδομένα για αυτά. Και σήμερα έχουμε ελάχιστα δεδομένα. Δεν ξέρω πόσο ποσοστό έχει χαρτογραφηθεί από το βυθό, αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Ε, και υπάρχουν παραδείγματα όπου ένα κράτος μέλος ε, έχει λάβει μέτρα προστασίας σε περιοχές όπου υπάρχουν ευαίσθητα είδη, ενώ ένα άλλο κράτος μέλος που βρίσκεται κήθεν των συνόρων δεν έχει κάνει το ίδιο πράγμα, οπότε πρέπει να φροντίσουμε να συντονίζονται όλα αυτά τα θέματα, είναι σημαντικό. Η χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας δεν είναι σημαντική μόνο προκειμένου περί της γαλάζιας ανάπτυξης, και της ε, εξερεύνησης ε, του πλούτου της σκήτης, αλλά όταν μιλάμε για προστασία των θαλάσσιων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χρειάζονται τα δεδομένα και πρέπει να τα έχουμε όλοι μαζί. Ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να υπάρχει μια υποχρεωτική μορφή για τα δεδομένα αυτά, ούτως ώστε να μπορούμε να τα συγκρίνουμε τα δεδομένα και θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ε, διάδοση των δεδομένων. Όλοι αναγνωρίζουμε νομίζω ότι είναι δημόσιος χώρος ο ωκεανός, οπότε το θέμα της εμπιστευτικότητας του εμπορικού απορρίτου επί των θεμάτων αυτών ε, συνοδεύονται από ένα ερωτηματικό και από την πλευρά μου είναι δημόσια ε, ιδιοκτησία, είναι η κληρονομιά των παιδιών μας, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται εκεί και με κάποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι ιδιοκτησία δημόσια. Πρέπει να είναι σαφές αυτό. Αυτό που είπε ο κύριος ε, Άνιου είναι επίσης πολύ σωστό ότι επιδοτούμε μεγάλα κομμάτια της κοινή αλλιευτικής πολιτικής προκειμένου περί συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και χτες ψηφίσαμε όπου πολλοί είπαν ότι πρέπει να επιδοτήσουμε κατασκευή νέων σκαφών και λοιπά, ναυπήγηση νέων σκαφών. Αν ε, ο κόσμος θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, τότε θα πρέπει και είναι λογικό να ζητήσουμε κάτι, ε, ένα αντίτιμο. Και νομίζω ότι η θέσπιση ε, της θάλασσας κοινού χώρου είναι το ελάχιστο, ελάχιστη προϋπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να της πω ότι συμφωνώ απολύτως με το έβρος αυτής ε, της εκθέσεως πρωτοβουλίας. Συζητήσαμε επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα θέματα αυτά και ε, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να πάρουμε αποφάσεις προσανατολισμού χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Διαφορετικά θα μπούμε σε ιδεολογικές συζητήσεις ε, ή διαφορετικά θα βρεθούμε ε, ε, απέναντι σε, μια γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος της πρόληψης ε, που βεβαίως θα οδηγούσε σε μια πλήρη παράλυση γιατί αν δεν έχουμε τα σωστά στοιχεία που είναι το α και το ω οποιασδήποτε πολιτικής θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε. Διαπιστώνουμε τα προβλήματα αυτά σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Πρώτον υπάρχουν αλλιευτικά αποθέματα τα οποία δεν ε, παρακολουθούνται επιστημονικώς, ιδίως στη Μεσόγειο. Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχει δυσκολία αξιολόγησης ε, της ε, υπεραλίευσης και έτσι ξεκινούν πολλές και δύσκολες συζητήσεις μεταξύ μας κυρίως όσον αφορά ε, την ε, ε, κατανομή της αλληλευτικής ικανότητας να και κράτος μέλους γιατί μια συνολική ικανότητα μπορούμε ενδεχομένως να την έχουμε. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, δεν έχουμε χαρτογράφηση του πυθμένα της θάλασσας και επομένως δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα πιο ευάλωτα σημεία αυτού. Επίσης αντιμετωπίσαμε ε, πρόβλημα παρόμοιο και σε άλλες περιπτώσεις ε, ε, και επομένως είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε αποφάσεις πολιτικές εάν δεν έχουμε την απαραίτητη γνώση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα δόκιμη αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας. Υπάρχουν και δύο άλλα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Ε, εξ αρχής να πω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες όσον αφορά δηλαδή, μια ιεράρχηση των δεδομένων, κυρίως όσον αφορά την ε, αλίευση και υπεραλίευση, γιατί είναι πολύ σημαντικό στόχο το θέμα της χαρτογράφησης ε, των, ε, του πυθμένα, καθώς επίσης και της καταχώρησης των πιο ευάλωτων σημείων, των αλλιευτικών πόρων που μπορούν να προχωρήσουν, που μπορούμε να διαμπορευτούμε, πολύ σημαντικό. και ε, διάφορα άλλα σημεία τα οποία δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε στη γενικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Ένα άλλο θέμα και το αναφέρατε πολύ στην έκθεσή σας, η εναρμόνιση των μορφοτύπων και της μεθοδολογίας έτσι ώστε και να υπάρχει δυνατότητα συγκρισιμότητας και να υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης στοιχείων. Ε, ε, δεν έχει καμία έννοια να έχουμε μία σειρά θαυμάσιων στοιχείων εάν δεν μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε και να τα ταξινομήσουμε ή να τα συγκρίνουμε. Ε, όσον αφορά τώρα τα όσα είπε ο Βρετανός συνάδελφος, νομίζω ότι το ερώτημα είναι άλλο. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μεγάλη Βρετανία, ναι ή όχι, αν ναι δεν υπάρχει ζήτημα το άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε, το οποίο ήδη σχετικά με τα, το κατά πόσον τα στοιχεία είναι δημόσια και αν θα πρέπει να υπάρχει απόρριτο, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος μεταξύ μας να δημιουργήσουμε μια ε, εσφαλμένη ε, ε, συζήτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ούτω ώστε τα στοιχεία και η ομαδοποίησή τους και η καταχώρησή τους να είναι προσβάσιμη σε όλου, επομένω, να είναι δημόσια στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό είναι άλλωστε και ο αντικειμενικό στόχος της δημοκρατίας. Πρέπει να είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Αντιθέτω, οι πηγέ μπορούν να καταχωρίζονται με τρόπον ώστε ε, να μην ε, υπάρχει ε, ειδική επίπτωση στους εμπορευόμενους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε μια εσφαλμένη συζήτηση πάνω στο ζήτημα αυτό, το οποίο μπορεί να το υπερβούμε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή ο κύριος Σέπαρτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι καλογραμμένη η έκθεση, δείχνει ότι η εισηγήτρια κατανοεί ε, καλά την κατάσταση όσον αφορά τα δεδομένα της αλληλείας. Ε, τα στοιχεία, όπως λέει, πρέπει να είναι ανοιχτά, αλλά ταυτόχρονα να καλύπτονται και από το απόλυτο, έτσι ώστε να διασφαλίζονται κάποια εμπορικά συμφέροντα μας ικανοποιεί. Θεωρούμε ότι γενικώ είναι μια καλή έκθεση. Αναφέρεται ότι τα αλλιευτικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα αφενός και συγκρίσιμα ε, με, με άλλα στοιχεία επίσης μας βρίσκει σύμφωνους ε, πρέπει ε, να υπάρχει δυνατότητα να ξεκινώντας από αυτά τα αλλιευτικά στοιχεία να φτάσουμε σε άλλα δεδομένα τα οποία θα μας δώσουν άλλες πληροφορίες που θα μας οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική αλληλεία ε, η Κομισιόν ε, θα μελετήσει ε, τις δυνατότητες που έχει έτσι ώστε να δοθεί συνέχεια στις στην έκθεση αυτή και βεβαίως ε, η έκθεση επιπτώσεων ε, θα είναι το τελευταίο στοιχείο, μπορεί ε, να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών και της βιομηχανίας και των θεσμικών οργάνων. Η επιχειρησιακή στόχη τώρα που θα ήταν να ενσωματωθούν όλες ε, οι ενωσιακές πρωτοβουλίες ε, για τα ε, θαλάσσια δεδομένα. Είναι αυτό που έχουμε κάνει ήδη και δηλαδή να ξέρουμε τι γίνεται στην, όσον αφορά την διαχείριση των θαλασσών, τον Κοπέρνικο κτλ. Ε, από την άλλη πλευρά να δούμε τι κάνει ο ιδιωτικός ε, τομέας έτσι ώστε να τους δώσουμε την δυνατότητα ε, να δώσουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία αλλά βεβαίω πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε όσον αφορά τη συλλογή αυτών των δεδομένων και κατά αυτή την έννοια θα συζητηθούν οι ενδεχόμενε επιλογέ που έχουμε. Τρίτος στόχος είναι να αναπτυχθεί μια καλύτερη ε, διεργασία βάσει της οποίας θα ε, ε, αποφασίζουμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται. Αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες δεν είναι σαφείς, ούτε είναι απολύτως σαφές που βρίσκονται τα μεγαλύτερα χάσματα ή δυσκολίες. Θα πρέπει να είμαστε είναι σχετικά εύκολο να αποφασίσει κανείς τις προτεραιότητες. Ε, δηλαδή, εάν ε, θέλει κανείς ε, να δει, ας πούμε, το βάθος του πυθμένα και θέλει το στοιχείο αυτό μόνο για την, για την εμπορική ναυτιλία, είναι πολύ εύκολο, αλλά εάν θέλει ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει το ίδιο στοιχείο ε, και για την βελτιστοποίηση της αλληλείας, τότε ενδεχομένως τα πρότυπα συλλογή θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Αυτοί είναι οι τρεις στόχοι λοιπόν της Κομισιόν ε, να μπουν όλοι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Κομισιόν σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Δεύτερον, να εμπλακεί περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας και τρίτον να αναπτυχθεί μια καλύτερη, ένας καλύτερος τρόπος επεξεργασίας έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση. Τώρα, ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής ε, ή υλοποίησης των στόχων ε, θα ε, διερευνηθεί μετά την μελέτη επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Eh, Κυρία Πατράνου Νέβες. Με βάση αυτά που άκουσα, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε κατά βάση. Το ζήτημα είναι σημαντικό. Η Αλία θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα της ε, διάθεσης των στοιχείων είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έγιναν και κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα ωφέλη μπορούν να προκύψουν ε, έγιναν δύο σχόλια προσθήκες οι οποίες, τα οποία ε, σχόλια τα έχω ήδη στην εκθέση απλά δεν σας το ανέφερα σε ό,τι αφορά την υπεραλίευση καταρχήν μιλάμε πάρα πολύ συχνά για την ε, υπερβολική ε, χωρητικότητα και δυναμικό, ικανότητα, λεπτική ικανότητα των σκαφών μας, αλλά με τρόπο πολύ ε, γενικό θα πρέπει να δούμε ε, για ποιο τύπου αλία υπάρχει γίνεται αλίευση, πού κλπ. Νομίζω ότι αυτό το project μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το πού ακριβώς και πώς ακριβώς γίνεται η υπεραλίευση ή υφίσταται η, η υπερβολική αλευτική ικανότητα. Και ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει ήδη στην έκθεση, απλά δεν το ανέφερα ε, επαρκώς και το σχολιάσατε, είναι η σημασία του project για τον προσδιορισμό των πιο ευάλωτων οικοσυστημάτων. Υπάρχουν βέβαια περιοχές οι οποίες έχει ήδη προχωρήσει πολύ χαρτογράφηση. Για παράδειγμα στην ε, αποκλειστική οικονομική στην, ε, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των νήσων Αζωρών. Εκεί έχει γίνει πολλή δουλειά. Έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί οι ευάλωτες περιοχές, αυτό πρέπει να το πούμε. Εγώ έχω ζητήσει ειδική προστασία για αυτές τις περιοχές που έχουν εντοπιστεί επιστημονικά, που έχουν οριοθετηθεί, ε, αλλά δεν, δεν υποστηρίχθηκα σε αυτό που ζήτησα. Συνεπώ α είμαστε συνεπεί. Πρέπει να γίνει δουλειά. Ένα από του στόχου είναι ο εντοπισμό των πιο ευάλωτων περιοχών, αλλά αυτή, αυτός ο προσδιορισμός, αυτή η ορθέτηση θα πρέπει να έχει και αποτελέσματα. Δηλαδή οριοθετούνται για να προστατευτούν κιόλα. Συνεπώ, α είμαστε συνεπεί. Όταν λέμε ότι είναι ευαίσθητοι σε αυτέ τι ζώνε, θα πρέπει αργότερα να υποστηρίζουμε και τι προτάσει προστασία του. Μετά, ετέθηκαν πολλά ζητήματα σχετικά με την διαθεσιμότητα των στοιχείων. Θα συμφωνήσω με την Ιζαμπέλ Τωμά που είπε ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε ένα ε, πρόβλημα εικονικό. Διότι αυτή τη στιγμή η τάση είναι η συλλογή των δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία απλώς δεν τα επεξεργαζόμαστε, δεν βρίσκονται σε ένα κοινό σημείο, ε, δεν τα έχουμε συλλέξει σε ένα κεντρικό σημείο. Οπότε αυτό που έχει ως στόχο η έκθεση είναι να ε, διευρυνθεί η συλλογή και η, διαθε... η... η θέση διαθεσιμότητα Η έκθεση λέει ότι αυτή η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να υπακούει ε, σε συγκεκριμένους κανόνες για το αν θα είναι επεξεργασμένα ή όχι στοιχεία με υποχρεωτική αναφορά στην πηγή έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να καταφύγουν εκεί για να ζητήσουν πιο λεπτομερή στοιχεία προσδιορίζουμε τη χρονική απόσταση ανάμεσα στην απόκτηση και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Αλλά αυτά τα διαφορετικά επίπεδα δεν έχουν σχέση με την απόκρυψη στοιχείων. Έχουν σχέση με την προώθησή τους. Τι εννοώ. Αν δεν καθορίσουμε διαφορετικά επίπεδα ε, δημοσιοποίηση των στοιχείων, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε ακόμα μεγαλύτερη απόκρυψη. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δοθούν κίνητρα. Αυτά δύο συνδέονται. Δεν πρόκειται να πετύχουμε την συλλογή μεγαλύτερης μεγαλύτερου όγκου χρήσιμων δεδομένων αν δεν έχουμε, δεν διαθέτουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτοί που συλλέγουν και κοινοποιούν αυτά τα δεδομένα έχουν, νιώθουν ότι έχουν κάτι να κερδίσουν. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας που θα λαμβάνει υπόψη τα κοινά συμφέροντα και θα οδηγεί στην δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό είναι το βασικό ερωτηματικό. Αν δεν καθορίσουμε διαφορετικά επίπεδα για διαφορετικούς τύπους δεδομένων και χωρίς κίνητρα, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην αποκτήσουμε καν αυτά τα στοιχεία. Ε, η, η, θάλασσα, όπως είπατε, είναι ε, δημόσια, δημόσιος χώρος, ναι, αλλά όχι μόνο η θάλασσα, και η γη και το διάστημα. Αλλά, όπως πολύ, πολύ συχνά έχω πει, και η χρηματοδότηση πολλές φορές είναι δημόσια και κρατική, Δεν θέλουμε να περιοριστούμε βέβαια στην δημόσια χρηματοδότηση, θέλουμε και την ιδιωτική χρηματοδότηση, αλλά επειδή ακριβώς η χρηματοδότηση ε, είναι και δημόσια και, για, και γίνεται το, το, το, το project υλοποιείται σε ένα κοινό δημόσιο χώρο, τότε υπάρχουν και υποχρεώσεις. Προκύπτουν, γι' αυτό το λόγο προκύπτουν και υποχρεώσεις. Ο στόχος πάντως είναι η βελτίωση της συλλογής και η διεύρυνση των δεδομένων που δημοσιοποιούνται. Αυτή είναι η πρότασή μου. Νομίζω ότι είναι ισόρροπη. Και θα βελτιωθεί με τις προτάσεις σας. Πατράου, οι τροπολογίε μπορούν να καταδεχθούν μέχρι τι 17 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Λέμε σημείο 13. Για μια ολοκληρωμένη αλληλευτική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στην περιοχή του Ειρηνικού, η γνωμοδότηση Πρωτοβουλία στι 29 Μαου ε, κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Συγγήτρια κυρία Φράγα, σήμερα θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Ο λόγος στην κυρία Φράγα καταρχήν και μετά στην Κομισιόν και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Κυρία Φράγα, το, το λόγο. Θα κάνω μια πιο σύντομη παρουσίαση σε σχέση με την άλλη φορά. Σας το είχα υποσχεθεί άλλωστε ότι δεύτερη φορά θα είμαι πιο συντομία. Ο δεύτερος λόγος βέβαια είναι ότι έχω βραχνιάσει, οπότε δεν νομίζω θα καταφέρω να μιλήσω 10 λεπτά. Ούτε 10 λεπτά. Την έχετε την έκθεση στα χέρια σας. Οπότε μπορείτε να τοποθετηθείτε επί ενός πολύ συγκεκριμένου κειμένου. Στόχος Τη της είναι ο καθορισμό μια αλληλευτική στρατηγική μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ε, ιδιαίτερο στον κεντρικό και δυτικό ειρηνικό σα είπα γιατί γιατί αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική ιδιαίτερα για τα τονοειδή 80% των ε, ε, ε παγκοσμίω ε, αυτού του είδους αυτής οικογένειας γίνονται εκεί, ε, αλλά είναι σημαντική και για άλλα είδη, μεταστευτικά είδη. Ταυτόχρονα αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ε, ενός αριθμού ε, νησιωτικών χωρών. Έχουμε 15 κράτη νησιωτικά Βανουάτου, Κυρμπάτη, νησί Μάρσαλ κλπ. Χαρακτηρίζεται πολύ, αυτή η περιοχή από παράνομη, άναρχη και μη καταγεγραμμένη αλία. Ενώ ταυτόχρονα ε, οι διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκλίνουν εκεί πολιτική, εμπορική πολιτική, πολιτική ανάπτυξης και αλληλευτική πολιτική τουλάχιστον. Η συμφωνία του Κοτονού ε, τελειώνει, εκπνέει το 2020 και τώρα εξετάζονται εναλλακτικέ λύσεις. Παρόλο που όλες αυτές οι λύσεις είναι διαφορετικές, έχουν περιφερειακή εστίαση. Γι' αυτό το λόγο μιλούμε για μια στρατηγική ε, μακροπρόθεσμη. Υπάρχουν ε, τρεις περιφερειακές οργανώσεις αλίας, η Διαμερικανική Επιτροπή ε, Τροπικού Τόνου καλύπτει την περιοχή από τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Χιλή. Έχουμε την Περιφερειακή ε, Οργάνωση, οργάνωση Αλίας του Ειρηνικού. Εδώ έχουμε οκτώ κυρίως ε, αλληλευτικά σκάφη και την οργάνωση αλίας του κεντρικού και νοτιοειρηνικού με τρία ε, ε, ε και 14 14 ε, στράτες. Είναι πολύ μικρή δηλαδή η ευρωπαϊκή παρουσία. Έχουμε συμφωνίες με το Κυριμπάτι της νήσου Σολομόντος και τη Μικρονησία. Η συμφωνία με τη Μικρονησία δεν έχει εφαρμοστεί. Ζητείται η πληρωμή του αντισταθμίσματος της προηγούμενης συμφωνίας. Η συμφωνία με τους νήσους Σολομόντος ε, επίσης έχει μπλοκαριστεί. Η μόνη που εφαρμόζεται είναι η Κυριμπάτη, η οποία μάλιστα θα ανανεωθεί. Η κυρία Λοβίν είναι η συγγήτρια για αυτήν την ανανέωση. Αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται λοιπόν από την ύπαρξη νησιωτικών κρατών κάτι που ε, δίδει στην ε, Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αντίθετα με άλλες περιφερειακές οργάνωσεις Αλίας, όπου τα, η μεγάλη πλειοψηφία των υδάτων είναι διεθνή εδώ έχουμε πολλές ΑΟΖ Μόνο 20% των υδάτων είναι διεθνή Και η αλία σε αυτά τα ύδατα δεν φτάνει ούτε στο 10% της συνολικής αλίας περιοχής. Τα ενδιαφέροντα λοιπόν των κρατησιωτικών αυτοκρατών είναι ιδιαίτερα αυξημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια στρατηγική πιο πολύ εστιασμένη στο κεντρικό και όχι στο δυτικό ειρηνικό. Γιατί η, ο κοινωτικό στόλο που βρίσκεται εκεί ε, έχει εστιαστεί. Βέβαια πιο πολύ στο Κυριμπάτι γιατί είναι πιο παλιά συμφωνία, αλλά τα συμφέροντά τους είναι αλλού. Γι' αυτό το λόγο ε, η, η Κομισιόν καταρχήν είχε ε, μάλλον η, η Κομισιόν είχε κάνει ένα λάθος και είχε εστιαστεί πιο πολύ στο δυτικό ειρηνικό, νήσι Σολομόντος κλπ. Εκεί που δεν λειτουργούν οι συμφωνίες, έκανε λάθος διότι τα συμφέροντά μας είναι στο κεντρικό ειρηνικό. Γι' αυτό το λόγο ε, η στρατηγική σχετικά με το, τις νήσους του Βάλου και Κουκ ε, στο κεντρικό ειρηνικό είναι πιο ενδιαφέρουσα θα μας ενημερώσει ελπίζω η Κομισιόν ε, διότι ε, έχουν, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για τις νήσους Κουκ ε, το, του Βάλου καθυστερεί λίγο περισσότερο βέβαια αλλά η εστίαση αυτή είναι πολύ καλύτερη στο κεντρικό ελληνικό Παραδοσιακά σε αυτή την περιοχή του ειρηνικού υπάρχει μια ένα ιστορικό ε, περιφερειακής οργάνωσης. Όπως σας είπα υπάρχουν ε, δύο οργανώσεις εκεί, ε, το Φόρουμ των Νησών του Ειρηνικού και το Φόρουμ η των Συμβαλωμένων Μερών της Συμφωνίας του Νουάρου. 14 εκατομμύρια δολάρια συν 4 εκατομμύρια πληρών οι είναι το ποσό στο οποίο έρχεται η συμφωνία που έχουμε υπογράψει ε, για τα 55 γρηγροί που ε, αλλιεύουν σε αυτήν την περιοχή πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα και την άλλη φορά είναι το σύστημα Vessel Day Scheme που χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες για την, τον έλεγχο της αλληλευτικής προσπάθειας. Είναι οι μέρες αλίας τις οποίες ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Το βασικό σύστημα, το βασικό πρόβλημα αυτού του συστήματος, το οποίο σύστημα δεν είναι κακό, αυτό καθ' αυτό, το οποίο όμως έχει επικριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους ε, είναι ότι, ε, θα, ότι είναι χρήσιμο μόνο αν γίνεται σεβαστό και είναι διαφανές. Ε, όμως δεν είναι σεβαστό, δεν γίνεται σεβαστό, οι ίδιοι δεν το σέβονται, θα το δείτε στον πίνακα που σας έχω αναφέρει. Αν στο μέλλον όμως εξασφαλιστεί αυτή η διαφάνεια, ναι, θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πτυχές, τις οποίες σας ανέφερα με μεγαλύτερες λεπτομέρειες προάλλες, να σας θυμίσω ότι υπάρχει ε, προσωρινή συμφωνία ε, σύνδεσης με την Παππούα και τα Φίτζη από το 2011 ε, για πρώτη φορά για μεταπημένα προϊόντα δόθηκε εξαίρεση, πλήρης εξαίρεση στους κανόνες προέλευσης εκείνη την εποχή ε, δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο, όχι μόνο στην, στην Ευρωπαϊκή Κοσερβοπία, που δεν είναι και τεράστια, που επηρεάζεται όμως, αλλά τις και τις επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτή η εξαίρεση σε τρίτες χώρες, που επίσης παράγουν κονσέρβες και διαθέτουν ένα σύστημα ειδικευμένων προτιμήσεων. Θα θυμάστε όσοι, πήγαμε στην, όσοι ήρθατε στις Σεϊχέλες ότι εκεί παραπονιόντουσαν για ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές οι εξαιρέσεις σε άλλες περιοχές όπως οι Σεϊχέλες ή και σε χώρες ε, ΑΚΕ. Όχι μόνο της χώρες του ειρηνικού. Συνεπώς, ίσως αυτές οι παραχωρήσεις ήταν υπερβολικές, αλλά να πω υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Τρέν ότι αντέδρασε και το πήρε πολύ στα σοβαρά τα πράγματα, γιατί είδε τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει το ζήτημα αυτό, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα χώρες Ακία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να αναδιαπραγματευτεί τη Συμφωνία Σύνδεσης σε όλη σε, όλες τις περιοχές, σε όλες τις χώρες και τις περιοχές για τις οποίες το θέμα της αλίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Γενική Διεύθυνση Trade σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μάρε κλπ. Σε συνεργασία μάλλον με τη Γενική Διεύθυνση Μάρε κλπ. Ε, προσπαθεί να διατηρηθούν αυτές οι παραχωρήσεις υπό την προπόθεση ότι και αυτές οι χώρες θα κάνουν παραχωρήσεις. Για παράδειγμα, να διευρυθεί να διευρυθούν αυτοί, αυτές οι εξαιρέσεις από τους κανόνες προέλευσης ε, όχι μόνο στα μεταποιημένα, να μην περιορίζονται μόνο στα μεταποιημένα αλλά και στα νοπά και σε αντιστάθμισμα ε, να μας ανοίξουν τα ύδατά τους αυτές οι χώρες σε δική μας ελευθερική προσπάθεια. Ε, από ό,τι ακούω, τα αιτήματα αυτών των κρατών ήταν υπερβολικά, συνέχιζαν να μην δίδουν εγγυήσει διαφάνειας, για παράδειγμα το Vessel Day Scheme κλπ. Οπότε από ό,τι άκουσα η συνεδρίαση μαζί του τελείωσε χωρίς αποτέλεσμα. Εντάξει, θα ξαναγίνουν και άλλοι γύροι διαπραγματεύσεων φαντάζομαι. Η έλλειψη διαφάνειας, όπως είπαμε, ε, δίνει λαβή σε ε, παρατυπίες. Για παράδειγμα, στο Βανουάτου και στις νήσους Φιτζή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί αυτές τις χώρες τρίτες χώρες μη συνεργαζόμενες σε ό,τι αφορά τον κανονισμό 1005 της ε, παρανομής άναρχης και μη δηλωμένης ε, αλίας. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά όλα αυτά είναι δεδομένα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη περισσότερη διαφάνεια στην διαχείριση της αλληλευτικής προσπάθειας. Το άρθρο 1 της Συμφωνίας Σύνδεσης ε, αναφέρεται στην βιωσιμότητα των ε, αλληλευτικών πόρων κλπ. Πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική τώρα. Με εξέπληξε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δεύτερη, ο δεύτερος σε μέγεθος δωρητή στον κόσμο μετά την Αυστραλία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στο δέκατο πρόγραμμα του ε, ε ταμείου, Ταμείου 745 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν ως βοήθεια συνολικά, μόνο το 2% για την αλία. Αυτό στο 10ο πρόγραμμα FED. Όμως, η αλληλευτική πορεία είναι από τους πιο σημαντικούς οικονομικά. Μόνο το 2% της αναπτυξιακής βοήθειας ε, του Ταμείου ε, Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγαν στην αλία. Από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος δωρητής στην περιοχή, οπότε Πώς είναι δυνατόν όλες αυτές οι χώρες να λένε ε, ότι η σημασία των ΗΠΑ και λοιπά είναι μεγαλύτερη. Γιατί, Γιατί παρόλο ότι δεν είναι ε, οι μεγαλύτεροι δωρητές γενικότερα αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά δίνουν περισσότερα χρήματα στην Αλία αυτές οι χώρες. Χιλή, ΗΠΑ, Πολιτείες, Αυστραλία κλπ. Σε αυτή την συνολική στρατηγική λοιπόν που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον σε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Είπα θα είμαι πιο σύντομα την άλλη φορά, αλλά τι, να πω. Θα, βελτιώσετε, θα βοηθήσετε να βελτιωθεί το κείμενο ε, τι προτείνω σε ε, βραχυπρόθεσμα, προτείνω να συνεχίσουμε με το Κυριμπάτι, με την, τον προσανατολισμό στο στην κεντρική ζώνη του ειρηνικού, να συνεχίσουμε με την καταπολέμηση της παρανομισαλίας και επίσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ε, EPA, ε, την ε, Συμφωνία εταιρική συμφωνία σύνδεση. Ε, θα δούμε, θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση να δούμε πού θα καταλήξει. Ε, μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μια πιο περιφερειακή προσέγγιση, να ακολουθηθεί μια πιο περιφερειακή προσέγγιση. Όπως και με όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια συμφωνία πλαίσιο, περιφερειακή συμφωνία πλαίσιο, ε, η οποία θα καθορίζει τις γενικές γραμμές της ε, αλευτικής μας δραστηριότητας εκεί στο μέλλον, τις, ε, τους δυνατότητες πρόσβασης, το, θέμα, θα καθορίζονται θέματα, θα θέματα διαφάνειας και διακυβέρνησης, καταπολέμηση της παρανομισαλίας και βέβαια τη συμφωνία, και εδώ συμφωνεί η κυρία Λεβέν, Ε, τη συμφωνία θα βασιστούμε στο VDS, ε, το Vessel Day Scheme, ε, αντί στην μέτρηση συγκεκριμένων ποσοτήτων αλλιευμάτων, ε, υπό την προπόθεση ότι αυτό θα γίνει πιο διαφανές. Αυτή, αυτό το, αυτή η συμφωνία πλαίσιο θα εξειδικευτεί βέβαια σε αναχώρα της περιοχής δεν έχει πολύ νόημα έτσι κι αλλιώς να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πολυμερή, δεν έχουμε τέτοια παρουσία με τα δικά μας τέσσερα γρηγοί, πώς να σε ανταγωνιστούμε τα 55 των ΗΠΑ για παράδειγμα. Ε, η αναπτυξιακή πολιτική επίσης θα πρέπει να παίξει σημαντικότερο και πιο δυναμικό ρόλο στην αλία. Τα νησιωτικά κράτη βέβαια δεν έχουν μεγάλες διοικητικές δυνατότητες. Ε, γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει η βοήθεια μας να διοχετευτεί μέσω της συνολικής βοήθειας, αναπτυσιακής βοήθειας που δίδεται σε αυτές τις χώρες. Ε, μια βοήθεια στον τομέα της αλίας από μόνη της δεν θα ήταν εύκολο να απορροφηθεί από τα κράτη αυτά. Αυτά την προηγούμενη φορά σας τα με περισσότερες λεπτομέρειες, οπότε νομίζω ότι μπορώ τώρα να αποσυρθώ και να σας επιστρέψω το μικρόφωνο. Merci Carmen. Tout le monde a bien compris que Carmen maîtrisait. Ευχαριστώ Κάρμεν. Η Κάρμεν παίζει στα δάχτυλα τον ειρηνικό και το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη διεξοδική έκθεση. Εν προκειμένου ε, έχουμε μια στρατηγική αλληλεία στον Ειρηνικό που έχουμε πολλά αλλιεύματα. Εκεί αυξάνεται η δραστηριότητα των ε, Ασιατών και καλά λέτε ότι υπάρχει μια ανισορροπία και ενδιαφέρεται η Ένωση να συνάψει αλλιευτικές συμφωνίες. Υπάρχουν πολλές που συζητούνται. Αναφέρθηκαν αυτές με χώρες Κυριμπάτη, ε, Νήσου, Σολομόντος, Μικρονησία. Στη Μικρονησία το υπέγραψε η Ένωση, εκείνοι δεν δέχτηκαν, το Κυριμπάτη συζητείται εντατικά. Η Ένωση θέλει να αρχίσει διαπραγματεύσεις και πολλές άλλες χώρες που δεν έχουν αρχίσει ακόμα διαπραγματεύσεις. Τώρα, πολλά είναι καλά από αυτά που είπε η συγγήτρια, θέλει περισσότερες συνέργειες, λέει ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των διαφόρων τομέων της πολιτικής, θα πρέπει να συνδυαστεί η πολιτική δράση και οι εξελίξεις και αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε γιατί η αναπτυξιακή πολιτική ε, πρέπει να ε, αναδειχθεί, το λέμε αυτό, πολιτική λοιπόν αλλίας και ανάπτυξης. Μετά η περιφερειακή εστίαση πρέπει να ενισχυθεί και αυτό πολύ σωστό, πολύ σημαντικό για την αλία την τοπική. Ε, διαφέρομαι λίγο σε σχέση με τη συμφωνία με το Κυριμπάτι, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που είναι υπέρ Άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί και εγώ είμαι μεταξύ των τελευταίων γιατί θεωρώ ότι ιδιαίτερα η περιφερειακή εστίαση είναι πολύ σημαντική για την αλληλιακή και η συμφωνία έτσι όπως είναι με το Κυριμπάτι δεν την στηρίζει, μάλλον το αντίθετο. Και πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι ακριβώς θέλουμε και πώς έχουν συνταχθεί οι συμφωνίες ώστε να επιδευχθούν οι στόχοι μας. Ε, τομεακή ε, υποστήριξη και αυτό είναι σημαντικό. Ε, χρειάζεται γι' αυτό το, ε, δημιουργία τοπικής αλίας, ε, πολύ σημαντική για τα κράτη εκεί. Τώρα αναρωτιέμαι αν πρέπει να υπάρξει υποδιέρεση στην βράχη και μέσο και μακροπρόθεσμη στρατηγική, διότι αν θέλουμε, που θέλουμε να φτάσουμε, κάνουμε ό,τι χρειάζεται από την αρχή. Στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις πρέπει να τονίσουμε πιο πολύ αυτό το θέμα των συνεργειών και να μην περιμένουμε αργότερα. Μπορεί να γίνει και νωρίτερα αυτό. Ή ζητούμε από την Κομισιόν να συνδέσει με τις χώρες και, και το ζήτημα της πρόσβασης. Αυτό καταρχήν είναι σωστό. Θέλουμε πρόσβαση να μην έχουν μόνο η Ασία και η ΙΠΑ, αλλά με ενδιαφέρει μια συνοχή στην αναπτυξιακή μας πολιτική και αυτό πρέπει να το τονίζουμε πάντοτε, ε, ιδιαίτερα όταν κάποια πράγματα ε, είχαμε ε, ανέκαθεν και πρέπει να αλλάξουν, όπως οι συμφωνίες αλληλείας παντού όπου συνάπτουμε συμφωνίες και έχουμε μια στρατηγική πρέπει να φροντίσουμε για τη βιώσιμη αλληλεία, να στηρίξουμε την τοπική αλληλεία και αυτό το λέει και η συγγήτρια. Χρειάζεται να δούμε σε ποιο βαθμό η τοπική αλληλεία μπορεί να προστατευτεί απέναντι στην παράνομη αλληλεία, γιατί έχουμε γιατί τα μικρά νησιωτικά κράτη έχουν περιορισμένους πόρους για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο, οπότε εδώ είναι αποφασιστική η συνεργασία μας μαζί τους. Είναι σημαντική η έκθεση όπως είπα, ιδιαίτερα επειδή η διμερής πολιτική ε, τονίζει την περιφερειακή διάσταση και ζητεί να συνυπολογίζονται και να συνεξετάζονται πολλοί τομείς πολιτικής ταυτόχρονα και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλα Λοβίν, ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση, επίκαιρη. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ΑΚΕ στον ειρηνικό πρόκειται να διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία εταιρική σχέση και η στρατηγική του ειρηνικού χρειάζεται στην Ένωση, χρειάζεται και η συζήτηση σχετικά. Ο ειρηνικός είναι από την στην άλλη άκρη του πλανήτη. Εγώ ε, είχα το προνόμιο να συμμετέχω σε κάποιες συναντήσεις μαζί με την κυρία Φράγκα και ήταν πολύ χρήσιμες οι συναντήσεις γιατί μπόρεσα να ακούσω επί τόπου τις συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τόνισε η κυρία Φράγκα ότι η Ένωση είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ε, δωρητής μετά την Αυστραλία αναπτυξιακής βοήθειας στην περιοχή όταν μιλάμε για δωρητές και η Ένωση ως αναπτυξιακός εταίρος έχει πολύ καλή φήμη στην περιοχή, αφού όλοι εκτιμούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που κάνει. Συμφωνώ με την κυρία Φράγκα απόλυτα ότι είναι περίεργο. Δεν το ξέρω εγώ ότι μόνο 2% της αναπτυξιακής βοήθειας πάει να στηρίξει την αλληλεία συμφωνώ ότι πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα, γιατί η βασική, ο βασικός φυσικός πόρος στην περιοχή είναι η αλία. Τα ψάρια έχουν. Έχουν το μεγαλύτερο απόθεμα τόνου στον κόσμο, 80% της παραγωγής τόνου προέρχεται σήμερα από τον ειρηνικό και τα περισσότερα βέβαια καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε ο βασικός καταναλωτής αυτού του τόνου. Υπάρχουν λοιπόν διασυνδέσεις εδώ μεταξύ της Ένωσης και της περιοχής του Ειρηνικού. Πρέπει βέβαια. Εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής, αλλά προκειμένου περί της αλίας έχουμε τέσσερα λιευτικά, 18 συνολικά, ε, τράτες, 14 τράτες βυθού. Δεν είναι πολλά και παραγάδι. Αυτά ε, είδα στις συναντήσεις που πήγα για την Ελία στην περιοχή, ότι υπάρχει μια ανισορροπία σχετικά με το πώς γίνεται αντιληπτή η Ένωση στην περιοχή. Γιατί μας έχουν πολύ ψηλά προκειμένου περί της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας και πολύ αρνητικά όταν πρόκειται για την Ελία. Γιατί να συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει διότι η Ένωση θεωρείται ότι δεν σέβεται τις περιφερειακές συμφωνίες για τη διαχείριση της αλίας και των αλλιευμάτων. Η Κομισιόν θα μας εξηγήσει βέβαια το περιφερειακό σύστημα, το VDS ε, που δεν είναι διαφανές κλπ. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το σύστημα που έχει ε, εγκαθιδρυθεί, θεσπιστεί από μικρές νησιωτικές ε, χώρες. Δεν θυμάμαι τώρα πότε έγινε αυτό, είναι κάποια χρόνια και αποδίδονται μέρες καφών ε, σε κάθε συμβαλόμενο μέρος και υπάρχει αυτό το σύστημα εμπορίας όπου μπορούν να κατανέμουν και να αγοράζουν, να εμπορεύονται μέρες. Τα, το σύστημα VDS το σέβονται και η Κίνα, η Αυστραλία, η Κορέα και η ΙΠΑ και όλοι. Τώρα οι τελευταία συνάπτουν νέα συμφωνία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, το κάνει αυτό. Ε, θέλαμε να έχουμε πρόσβαση με βάση το ίδιο σύστημα, ε, το τονάζ δηλαδή, το οποίο ίσχυε σε ελληνικές συμφωνίες. Και αυτό δημιούργησε μεγάλες εντάσεις στην περιοχή και η κυρία Φράγκα μπορεί να το βεβαιώσει αυτό. Ακούμε τους εκπροσώπους των μικρών νησιωτικών κρατών να λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φύγετε. Δεν μπορεί να έρχεστε και να μας επιβάλλετε εσείς τι θα κάνουμε. Οπότε όλα αυτά δημιουργήσαν μεγάλες εντάσεις. Και όταν πρόκειται για το, τη Συμφωνία Κυριμπάτη, αυτό θα το συζητήσουμε περισσότερο αργότερα, στα πλαίσια της δικής μου της έκθεσης. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κυριμπάτι διαπραγματεύτηκαν μία συμφωνία που υπεγράφει από το Κυριμπάτι αλλά είναι εκτός από το σύστημα VDS και αυτό δημιούργησε πάρα πολλές συζητήσεις στην περιοχή και δημιούργησε οργή και επιθετικότητα επίσης προς, ε, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπε ήδη η κυρία Φράγκα, οι νήσεις Σολομών και η Μικρονησία και οι δυο αρνήθηκαν να επικυρώσουν συμφωνίες με την Ένωση ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή λένε ότι δεν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρχεται και να μας λέει πώς θα κάνουμε εμείς διαχείριση των συστημάτων, εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το σύστημα VDS και εσείς μας λέτε να μην το εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι επικοδομητικός εταίρος στην περιοχή. Δηλαδή χρησιμοποιώντας την αναπτυξιακή βοήθεια για να στηρίξει τα μικρά νησιωτικά κράτη στην ανάπτυξη, να εφαρμόσει τη συμφωνία για τα μέτρα του κράτους λιμένα, να βοηθήσει στην καταπολέμηση της άναρχης παράνομης αλίας, λαθραίας αλίας, πλά. Να βοηθήσει σε επιστημονικά θέματα στη συλλογή των δεδομένων. Σε όλα αυτά μπορεί να είναι επικοδομητικός εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσει και μια θετική εικόνα στην περιοχή υπέρ ότι δηλαδή συνεργαζόμαστε εμείς. Αυτό το χρειαζόμαστε και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να το εξασφαλίσουμε όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις για το EPA, την Συμφωνία Εταιρικής Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρείται ως ένας εταίρος που πάει εκεί για να αρπάξει τους αλληλευτικούς πόρους και να τους πει και τι θα κάνουν. Είμαστε ε, από τους μεγαλύτερους δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας και πρέπει να προσέχουμε πολύ την εικόνα μας, την εικόνα που προβάλλουμε στην περιοχή. Κατόπιν τούτου, η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης και η κυρία Φράγκα τώρα προτείνει να μην δώσουμε ε, παρεκκλήσεις στους κανόνες καταγωγής σε άλλα νησιωτικά κράτη, εκτός και αν μας εξασφαλίσουν και εκείνη την πρόσβαση στην Αλία. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου της κυρίας Φράγκα. Α, είναι η πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Μου φάνηκε ότι το διάβασα σε δικό σας, στο δικό σας κείμενο. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Φράγκα. Η κυρία Φράγκα λέει ότι δεν είναι η δικιά της πρόταση αυτή, είναι η πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Αλλά στο σημείο 11 στην έκθεση λέει ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να δώσει άλλες παρεκκλήσεις εκτό εκτός από αυτούς που έχουν διαπραγματευτεί ε, αν δεν υπάρξει ε, αμοιβαίο όφελος για την ευρωπαϊκή αλληλεία όπως πρόσβαση στους ελευτικούς πόρους ε, μέσα στην ΑΟΣ αυτής της χώρας. Είναι το σημείο 11 της έκθεσης. Ε, μπορώ να το απευθύνω αυτό και στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, γιατί θα, θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πολύ ευαίσθητοι στι διαπραγματεύσει. Γιατί οι συμφωνίε εταιρική σχέση, από ό,τι κατάλαβα και από την πλευρά τη ομάδα των Πρασίνων, θα πρέπει να είναι μια πραγματική εταιρική σχέση και ένα αναπτυξιακό μάλλον παρά εμπορικό εργαλείο. Εμείς έχουμε ένα χρέος προς τις χώρες αυτές που ήταν κάποιες από αυτές απικίες ευρωπαϊκών χωρών, τώρα είναι αναπτυσσόμενες χώρες, οπότε ο βασικός στόχος μιας οικονομικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης πρέπει να είναι η συνεργασία, η υποστήριξη και η ανάπτυξη. Δηλώνω ότι η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτό το θέμα του πώς θα ζητήσουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να μας αφήσουν να ε, μπούμε στο βασικό τους φυσικό πόρο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη αγορά, με μεγάλη ισχύ, είναι μεγάλος δωρητής, μπορεί να δοθεί η εντύπωση ότι πάμε να τους ε, πιέσουμε και να τους εξαναγκάσουμε και να τους πούμε δώστε τα ψάρια, αλλιώς δεν θα σας εξασφαλίσουμε πρόσβαση στις αγορές μας είναι πολύ λεπτή. Λεπτές ισορροπίες είναι αυτές και πρέπει να τις ε, σεβαστούμε. Τέλος, να ρωτήσω την κυρία Φράγκα κάτι για την παρέκκληση από τους κανόνες καταγωγής, γιατί εκφράζεται πολλές ανησυχίες σχετικά με την νομοθεσία απλά και ότι πολλές χώρες μπορεί να θέλουν να παρακάμψουν την νομοθεσία απλά ε, και να μην τη βάλουν την νομοθεσία αυτή στην ε, συμφωνία. Μπορεί να το κάνουν αυτό. Μήπως ε, η Κομισιόν εδώ θα πρέπει να αντιδράσει και να το φροντίσει αυτό το θέμα. ε, τώρα για την υπέρβαση των ημερών των σκαφών. Θέλω να, πω, να το πω αυτό γιατί ήδη στο Κυριμπάτι έχουν υπέρβαση κατά πάνω από 80% των ημερών των σκαφών και αυτό είναι μια ηρωνία δεδομένου ότι είναι χώρα με την οποία έχουμε συμφωνία, οπότε δύσκολα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει να τους πει ότι εμείς επικρίνουμε το VDS ενώ έχουμε συμφωνία με εκείνη τη χώρα που έχει τη μεγαλύτερη υπέρβαση στο, στις ημέρες των σκαφών στα πλαίσια του VDS. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο ε, Σεζαρή από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Καταρχήν ε, χαιρετίζουμε θερμότατα την έκθεση αυτή για τον ειρηνικό και ευχαριστούμε την εισηγήτρια που έθεσε το θέμα αυτό με τρόπο που απηχεί την ανακοίνωση της Κομισιόν για την συνεκτικότητα της πολιτικής μεταξύ αλληλείας, εμπορίου, περιβάλλοντος και οπωσδήποτε αυτό μπορεί να το δούμε ως ένα παράδειγμα περιφερειακής προσέγγισης που περιλαμβάνει μεγαλύτερο συντονισμό, συνεργασία και συνοχή, όπως είπα, όχι μόνο μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν, αλλά και μεταξύ των πολιτικών. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι βρίσκουμε πολλά στοιχεία τα οποία επιδιώκαμε μέσα από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εξωτερική διάσταση, θέματα όμως που περιλαμβάνονται και στην έκθεση της κυρίας Λουβέν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη ανακοίνωση της Κομισιόν και εντοπίσαμε το, το βασικό στοιχείο εδώ που είναι η ανάγκη να υπάρχει συνεκτική, κοινή, επιμερισμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομέων, αλληλή, ανάπτυξη, εμπορίου. Τώρα, ποιο είναι το σημείο κινήσεώς μας, όποιος και αν είναι ο τομέας, η πολιτική. Ε, το σημείο κινήσεως είναι η βιωσιμότητα η διατηρησιμότητα. Και αυτό κάνουμε στην πολυμερή δράση, ε, στα FPA, στα EPA, στις διάφορες συμφωνίες μας. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση αυτή. Και έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα έτσι, ε, αυξημένη ε, συνοχή και συνεκτικότητα. Η βιωσιμότητα σημαίνει διαχείριση των πόρων προφανώς, αλλά και καταπολέμηση της πλά, παράνομη λαθρέα αναρχιαλία, πολιτική ελέγχου και οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να έχουμε ένα πολυμερές σύστημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για πολύ μεταναστευτικά είδη. Το 90% των αλλιευμάτων αυτών των πολύ από ε, μεταναστευτικών ειδών είναι στην ΑΟΖ υπάρχει ένας πολυμερής οργανισμός που διαχειρίζεται ε, συνολικά αυτούς τους πόρους. Χωρίς την πολυμερή συνεργασία λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα στη διατήρηση των πόρων. Περιφερειακή προσέγγιση λοιπόν, ε, όπως προβλέπετε και στην έκθεση αυτή, είναι ακριβώς ο στόχος μας στην WCSP και στις εταιρικές σχέσεις. Μπορούμε να πούμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουμε να μας βλέπουν, όπως είπε και η κυρία Λοβέν, ως ο καλύτερος φίλος, ένας επιστήθιος φίλος, αλλά μπορώ να εξηγήσω γιατί δεν μας βλέπουν επιστήθιους φίλους. Εμείς δεν είμαστε πολύ ευτυχείς με το σύστημα αυτό το VDS για συγκεκριμένο λόγο. Το VDS δεν επιτυγχάνει τον στόχο που αξίωναν ότι θα εξυπηρετούσε. Και είναι και θέμα αριθμών. Αυτό το πρόγραμμα ίσχυσε για πρώτη φορά το 2008. Ήταν ένα μέτρο που υπήρχε τότε. Τότε υπήρχε πάγωμα των ημερών, ήταν περίπου 30.000 ημέρες και όταν το αναλύσαμε το 2011, λίγα χρόνια μετά, τι συνέβη. Οι μέρες ε, που αναφέρονταν στον αρμόδιο φορέα ήταν 46.000 και αυτές οι μέρες ε, ε, είναι αλληλεία κυρίως στην ΑΟΖ. Οπότε η ευθύνη τους ως κράτος που, αλληλευτικό είναι να φροντίσει ότι θα έχει παρουσία ανάλογη με άλλες περιοχές του κόσμου και στη Βόρεια Θάλασσα έχουν ληφθεί μέτρα που δεν μας ε, ικανοποιούν απόλυτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να πει αυτό που πιστεύουμε για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Αν δεν είναι πράγματα που τους αρέσουν ή αν ε, ακούν διαφορετικά πράγματα από ότι όταν συζητούμε για το Ταμείο Ανάπτυξης, και τα κονδύλια ανάπτυξη, τι να κάνουμε. Αυτά πιστεύουμε για την Ελία. Σε ό,τι αφορά την μέσο και βράχη πρόθεσμη προσέγγιση, εμεί πιστεύουμε ότι είναι καλή. Γιατί σίγουρα μια περιφερειακή προσέγγιση και με την ενδεχόμενη συζήτηση και ενδεχομένε μελλοντικέ διαπραγματεύσεις με το FFA, ε, είναι καλή ιδέα. Αλλά θα είναι μακρές και περίπλοκες αυτές οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και δεν πρέπει και εδώ να ξεχνάμε ότι δεν είναι ε, όλα τα FFA ικανοποιημένα από το σύστημα VDS το οποίο εφαρμόζονται ε, από, όχι από την FFA αλλά από την Συμφωνία του Ναουρού. Βράχει πρόθεσμα όπως αναφέρθηκε ε, ίσως αυτές τις μέρες θα πάρουμε από το Συμβούλιο την εντολή για να αρχίσουμε επίσημα διαπραγματεύσεις για βιώσιμες συμφωνίες με τις νήσους Κουκ. Οπότε θα αρχίσουν επίσημες διαπραγματεύσεις ε, τη βδομάδα που θα αρχίσει 22 Ιουλίου και οι διαπραγματεύσεις και η εντολή από το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει επακριβώς τις αρχές που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Δεν θα παρεκκλίνουμε δηλαδή από αυτή τη γραμμή. Η ό,τι αφορά τώρα της, ΕΠΑ, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, έχει επιτύχει αρκετά, συνεργαζόμαστε μαζί τους για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και αν το σύστημα, όπως είπαμε στην WCPFC, δεν συνιστά πρόβλημα καταρχήν, γιατί δεν είναι ότι έχουμε αντίρρηση στο σύστημα καθ' αυτό, αλλά το σύστημα δεν είναι διαφανές. Και για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα και εγώ όλα αυτά τα δεδομένα που ανέφερε η κυρία Λοβίνη, γιατί έχω πάει τρεις φορές ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας και δεν έχω καταλάβει πόσες μέρες χρησιμοποίησαν οι στόλοι από την Ασία και την, ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε μέχρι την επαναδιαπραγμάτευση. Γιατί μέχρι πέρσι είχαν αποκλειστεί από το VDS σύστημα. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που πλήττει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πω ότι Έχουμε τέσσερα γρηγρή και τέσσερα παρα... Ε, ε, λιευτικά με παραγάδι, όχι δεκατέσσερα. Ε, υπάρχει δυνατότητα αλληλείας ε, ξηφία, αλλά τα ενεργά ήταν τέσσερα-πέντε το πολύ με παραγάδι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν μπορεί να θεωρείται κύρια απειλή για τη βιωσιμότητα εκεί. Από την άλλη πλευρά θέλουμε να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα. Πράγμα όχι πάντα εύκολο, όπως ε, είπαμε στις συζητήσεις ε, με τους Αμερικανούς και τους ε, Ασιάτες εταίρους μας. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες για τα διάφορα FPAs, αλλά θέλουμε συνεκτική προσέγγιση πάντως στα διάφορα FPA τις διαπραγματεύσεις. Γεωγραφικά η Μικρονησία και η νήσι Σολομών δεν είναι το κύριο μέλημά μας, ε, αλλά ε, και εκεί υπάρχουν μεταναστευτικά είδη, οπότε οι στόλοι εκείνη την εποχή ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τα αποθέματα. Η νήσι Κουκ είναι σε πιο κεντρική θέση και ε, είναι πιο πολύ κοντά στη στρατηγική μας, αλλά είναι χώρα αγοράς Θέλουμε λοιπόν ε, να γίνεται βιώσιμη αλία εκεί. Και από ό,τι καταλάβαμε από τις λίγες πληροφορίες που μας έδωσαν ε, οι φίλοι μας από τις μικρές νησιωτικές περιοχές, αυτό το σύστημα το δεν είναι ε, σαφές, το VDS δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικό και θέλουμε βεβαίως ε, διευκρινήσεις για να μπούμε και εμείς στο σύστημα και σε μέρες. Γιατί να μην υπάρχει ε, παντού ένα σύστημα VDS, αλλά με προϋπόθεση ότι θα είναι σαφές, διαφανές και θα μπορεί να γίνει ε, κατανοητό από τον κόσμο. Ευχαριστώ κυρία, κύριε Σεζαρή για τις επεξηγήσεις και διευθύνσεις που μας δώσατε. Ο ειρηνικός είναι μεγάλος ε, και ευρύς. Για να ολοκληρώσουμε, σύντομα Κάρμεν, σε παρακαλώ. Να πω στην κυρία Λοβίν ότι και η ίδια υποπίπτει σε αντιφάσεις. Μου λέει ότι το κυριμπάτι ε, δεν σέβεται το σύστημα Vessel Day Scheme. Ίσως, λοιπόν, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε μια συμφωνία με βάση το βάρος. Οπότε η ίδια αναγνωρίζει ότι το vessel skin δεν τηρείται, δεν τιμωρούνται όσοι το παραβαίνουν, δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, διότι όπως είπε και η Κομισιόν, κανένας δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί. Επιπλέον όμως, η συμφωνία του vessel skin, η συμφωνία του Παλάου δηλαδή, έχει μια υποσυμφωνία αυτή της μικρονησίας η οποία αναφέρει πως το σύστημα Vessel Day Scheme εφαρμόζεται για τις χώρες της συμφωνίας του Ναούρου για την μεταξύ τους ανταλλαγή ημερών αλίας. Συνεπώς το Vessel Day Scheme εφαρμόζεται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αλίας ε, κατά το δοκούν. Ο μόνο τους για παράδειγμα ε, αποφάσισαν να το χρησιμοποιήσουν που δεν ε, λεωποιήθηκε η συμφωνία τελικά και το κρυμπάτι δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Κομισιόν δεν το προτιμάει, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα της αλίας με βάση αυτό το σύστημα. Στην Πολυμερή Συμφωνία των ΗΠΑ, για παράδειγμα, το Vessel Day Scheme δεν εφαρμόζεται. Υπάρχουν κάποιες ονομαστικές θεωρητικές μέρες, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στην τελευταία έκθεση για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης αναφέρεται ότι το 2011 η ε, ονομαστικές ημέρες των ΗΠΑ ήταν 2.770 και οι πραγματικές ημέρες αλίευσης αλίας ήταν 8.000. Συνεπώς δεν εφαρμόζεται ούτε με τις ΗΠΑ το Vessel Day Scheme. Από την άλλη μεριά, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόσωπος της Κομισιόν, στην Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας υπάρχουν χώρες, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αμφισβητούν το VDS δεν δίδεται καν σαφής ορισμός του τι είναι η μέρα αλίας. Διότι η μέρα αλίας ε, εξαρτάται, ε, ε, συναρτάται από το μήκος του σκάφους κλπ. Και άλλους παράγοντες. Για αυτούς, για αυτές τις χώρες το σύστημα αυτό αποτελεί απλώς ένα πρόσχημα για να εισπράττουν ποσά. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι, αλλά αυτό κάνουν. δεν το σέβονται ούτε οι ίδιες οι χώρες αυτό το σύστημα. Πολύ δε περισσότερο που μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά μπορεί και να μην εφαρμοστεί για ξένους τόλους. Το Κυριμπάτι δεν το εφαρμόζει. Σε ό,τι αφορά την Συμφωνία Σύνδεσης, την υποστηρίζω υποστηρίζω την Κομισιόν που το διαπραγματεύεται. Γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις ε, τελωνιακές ε, ε, παραχωρήσεις για να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη τρίτων χωρών. Και προφανώς τα προϊόντα θα πρέπει να είναι τοπικής παραγωγής προκειμένου η χώρα να εποφεληθεί του συστήματο αυτού. Ε, Προφανώ, διότι αν εγώ υπάρχω μια σύμφωνα με την Νέα Γουινέα, θα πρέπει τα προϊόντα να προέρχονται από την Νέα Γουινέα, όχι από την Ταϊλάνδη, γιατί αλλιώ ε, δεν ενθαρρύνω την παραγωγή τη Νέα Γουινέα, αλλά την παραγωγή τη ε, Ταϊλάνδη και του στόλου άλλων χωρών. Αυτό συμβαίνει με την παγκόσμια Νέα Γουινέα. Οι Φιλιππίνε και η Ταϊλάνδη ε, πάνε εκεί, ε, ε, επενδύουν για να εποφεληθούν του συστήματος ε, των, ε, του πρωτομισιακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, συμφωνώ με την Γενική Διεύθυνση Trade. Αν θέλουμε να διευρυνθεί αυτή η παρέκκληση των, από τους κανόνες προέλευσης, που δεν συμφωνώ να γίνει έτσι, να γενικευθεί αυτή η παρέκκληση, γιατί θα ε, εποφελθούν και άλλες τρίτες χώρες, θα πρέπει να, προχωρήσουμε, να προσέξουμε. Αν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο πάντως, να πούμε, να το μελετήσουμε, αλλά κάτι θα πρέπει να παραχωρήσετε κι εσείς. Δεν είναι δυνατόν εμείς να χρηματοδοτούμε την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες. Οπότε θα πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά τα πράγματα. Μετά, σε ό,τι αφορά την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Συμφωνώ γιατί αξιολογούν τόσο θετικά την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά, αλλά όχι στην τομέα της Αλία. Γιατί η αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα της Αλία είναι πολύ μικρή. Δεν πρόκειται μόνο για ενίσχυση στην τοπική αλία, για τα, στα τοπικά λευτικά σκάφη κλπ. Πρόκειται και για βοήθεια στην υποδομή, στα λιμάνια κλπ. που δεν δίνεται αυτή τη στιγμή. Θα, έκανε, θα τους έκανε όλους πολύ πιο πλούσιους αν διδόταν. Γιατί σε αυτές τις χώρες υπάρχει έλλειψη υποδομών. Τα σκάφη μας, τα σκάφη τα αμερικανικά, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καν υποδομέ διότι δεν υπάρχουν υποδομέ. Ωραία, εντάξει, το βουλώνω, κατάλαβα. Ναι, είναι πολύ ωραία που σε συνεπέρνει το πάθο σου, Κάρμεν. Λοιπόν, κατάθεση τροπολογιών 18 ε, Ιουλίου και 5 Σεπτεμβρίου ψήφισε στην Ολομέλεια. Στην ε, Επιτροπή, συγγνώμη. Ευχαριστούμε για αυτήν την ε, πλούσια και επικοδομητική συζήτηση. Θα περάσουμε τώρα στην τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κινητικού συστήματος ελέγχου τη στήριξης των κανόνων κοινή αλληλευτικής Πολιτική. Ε, πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα γιατί αφορά τον έλεγχο. Η συγγήτρια είναι η Ιζαμπέλ Τομά και θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Ιζαμπέλ Τομά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο εργασίας, όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, δεν είναι προέκθεση, απλώς ένα έγγραφο μεθοδολογίας ε, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε σε ποια <clears throat> μία συμφωνούμε όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ε, θα προχωρήσουμε σχετικά ε, με την διαδικασία ε, ε, θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Στην ουσία πρόκειται για την ταξινόμηση των διαφόρων μέτρων του κανονισμού ελέγχου σε δύο κατηγορίες από ό,τι λέμε συνήθως, αλλά, συνήθως, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις είναι οι εφαρμοστικές πράξεις, η κατεξουσιοδότηση και η συναπόφαση. Γιατί προτείνω αυτό το μεθοδολογικό προέγγραφο, διότι θεώρησα ότι κινούμεθα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, δηλαδή τον τομέα του ελέγχου. Ε, έχουμε περίπου 60 μέτρα ε, κανονισμού ε, τα οποία τουλάχιστον ορισμένα μεταξύ αυτών είναι πολύ ευαίσθητα και από τα οποία προκύπτουν κυρώσεις κυρίως όσον αφορά την ανέρεση των αδειών ας πούμε, η αναστολή αδειών και οτιδήποτε σχετίζεται με ενδεχόμενη κύρωση θα πρέπει ε, λόγω της ευαισθησίας του να ελέγχεται ε, και από τον κλάδο αλλά και από τους απλούς ε, πολίτες. Θα επανέλθω σε αυτό. Είναι γεγονός πάντως ότι το θέμα της υπόνοιας, της δυσπιστίας που έχουν ε, οι επαγγελματίες για το τι συμβαίνει στη διπλανή χώρα, τι γίνεται στη διπλανή και τι έλεγχοι γίνονται και η δυσπιστία που συχνά δείχνουν οι πολίτες όσον αφορά τους ελέγχους μας κάνει πιο προσεκτικούς. Πάντα όσον αφορά τη μεθοδολογία βεβαίως εμείς ε, πρέπει, αυτός είναι ο ρόλος μας, ε, να προωθήσουμε τις αποφάσεις προς ένα από τα τρία, τρεις επιλογές ε, που σας ανέφερα προηγουμένως ε, σε συνεργασία βέβαια και με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, δηλαδή του Συμβουλίου. Έχουμε ε, της ε, κατεξουσιοδότηση ε, πράξης. Εδώ γίνεται η επιλογή με ε, εκ των υστέρων έλεγχο του Κοινοβουλίου, αλλά από την άλλη πλευρά ε, μπορούμε να κρατήσουμε μια σειρά από αυτά τα μέτρα ε, στην στη συναπόφαση. Κάνω λοιπόν δύο προτάσεις. Η πρώτη αποσαφηνίζω μάλλον να το πω διαφορετικά ορισμένες από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις έτσι, ε, πράξεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στα έγγραφα της Κομισιόν θα μπορούσαν οπωσδήποτε άνετα να περάσουν σε εφαρμοστικές και ε, το αντίστοιχο μπορεί επίσης να γίνει και ε, να καταλήξουν τελικά οι μεν και οι δε στην απόφαση. Από νομική άποψη μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μάλλον ιεράρχηση ε, και ε, πολιτική πράξη στην ουσία. Μπορεί να είναι πολιτική απολύτωση στην απόφαση και μετά σιγά σιγά κατεβαίνουμε σε κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικές ε, πράξεις. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια μεγάλη γκρίζα ζώνη η οποία παραμένει έτσι αχαρτογράφητη και η οποία χρήζει οπωσδήποτε αντιμετωπίσεως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η πρόταση λοιπόν είναι να προχωρήσουμε σε κάποια ιεράρχηση ανάμεσα στο πιο εκτελεστικό ε, επίπεδο και το πιο πολιτικό επίπεδο αντιστοίχως, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δοθούν και παραδείγματα, να δοθούν και ιδέες περί ποιου επίπεδου μιλάμε. Ας πούμε, ε, η ε, μεθοδολογία για, τις, για την εκφόρτωση ε, θα μου πείτε ναι, είναι ε, εκτελεστικές πράξεις. Ναι, αλλά εάν αποφασιστεί, ας πούμε, και άλλωστε το συζητήσαμε προηγουμένως ε, με την έκθεση πρωτοβουλία της κυρίας Πατράου Νάβες. Εάν αποφασίσουμε ότι ε, η μεθοδολογία διασάφησης θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως έτσι ώστε ε, να έχουμε τη δυνατότητα χρήσης και ομαδοποίησης των στοιχείων και επομένως να πούμε ότι θα έχουμε ένα έγγραφο ενιαίο για αυτήν την διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που στην αρχή φαίνεται απλό τελικά εξαρτάται από αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, αυτό που αποφασίζουμε να κάνουμε. Το ίδιο ισχύει ε, και με το εάν αποφασίσουμε να έχουμε συστήματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρονικής καταχώρησης, εάν θέλουμε να έχουμε ε, πληροφορίες αυτής ε, της καταχώρησης, ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο να έχουμε συστήματα συνεκτικά και συγκρίσιμα, έτσι ώστε η σύνδεση να μπορεί να γίνει εύκολα και αποτελεσματικά. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, έστω και αν το ζήτημα είναι να υπάρχει σωστή ιεράρχηση των δικών μας ε, είδη προσανατολισμών, υπάρχει και ε, μία δεύτερη τροχιά εργασίας την οποία σας προτείνω. Η ιεράρχηση της ε, εναρμόνισης, αλλά είναι πιο ευαίσθητο το θέμα όταν μιλάμε για τον έλεγχο, ο έλεγχος απαιτεί μεγαλύτερη εναρμόνιση έτσι ώστε να αποφευχθεί η δυσπιστία και η καχυποψία από πλευράς ε, των ε, επαγγελματικών του κλάδου που πάντα πιστεύουν ότι οι έλεγχοι δικοί τους είναι περισσότεροι από ότι τον, στους γειτονές τους, στο γειτονικό κράτος και των πολιτών που πιστεύουν ε, ότι οι έλεγχοι που γίνονται στην αλληλεία συχνά δεν είναι ε, αυστηρή. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Επίσης, ε, να επαναλάβω ότι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ε, κυρώσεις χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία. Για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εδώ μια σημαντική ευκαιρία με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, κυρίως ε, την ε, ευκαιρία να δηλώσει εξ αρχής το περιεχόμενο του εκτονιστέρων ελέγχου προς τις κατεξουσιώδες πράξεις. Ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε στις αιτιολογικές του σκέψεις να δηλώσει ότι στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ασφάλεια ε, ή με τα δεδομένα ε, για α, β, γ λόγους ε, θα αφορούν περισσότερο κατεξουσιοδότηση και όχι εφαρμοστικές πράξεις, έτσι ώστε να προσανατολιστεί καλύτερα η εργασία της Κομισιόν στον τρόπο με τον οποίο ε, θα αντιμετωπίσει τις, τα μέτρα αυτά. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα ενός κατά κάποιο τρόπο προσχεδιασμού, πρώιμου σχεδιασμού βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας προσχεδιασμού, λέω, του ελέγχου που η συνθήκη της Λισαβόνας ε, δίνει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να κάνει εκ των υστέρων. έτσι ώστε ε, να μην υπάρχει και εκ των υστέρων συχνή αμφισβήτηση των κατεξουσιώδης πράξεων έτσι όπως έχουν ληφθεί από το Κοινοβούλιο. Έχουμε άλλωστε και την έκθεση Σάντσες Πρεσέντο που αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα να κάνει αυτόν τον εκ των έλεγχο ε, με τα μέσα τα οποία θα αποφασίσει να δώσει στον εαυτό του. Όσον αφορά τους εκτονιστέρων ελέγχους λοιπόν, καλό θα ήταν να έχουμε την δυνατότητα ήδη ε, μια και μιλάμε για κανονισμούς ελέγχου, να αφήσουμε, να δώσουμε μια ιδέα ε, έτσι ώστε να προειδράσουμε και την Κομισιόν για το ποιες θα είναι οι θέσεις μας. Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Τομάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είχα την ευκαιρία να διαβάσω την ε, ε, πρώτη αυτή το προσχέδιο έκθεσης και συμφωνώ με τη θέση της εισηγητρίας. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου από τη μία πλευρά την αναμόνηση και από την άλλη μεριά την δικαιοσύνη. Ε, την ε, ισοδικία γιατί ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα πολύ σαφές μήνυμα έτσι ώστε να μην καταλαβαίνουν, να μην κατανοούν, να μην αντιλαμβάνονται τα μέτρα και τους κανόνες με διαφορετικό τρόπο οι διάφορες χώρες. Νομίζω ότι αυτά είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, έχουμε την γνωμοδότηση της ε, ε, ΛΥΜΠΕ. Βέβαια πολύ συχνά το πρόβλημα όπως ξέρετε δεν είναι ο ίδιος το ίδιο το νομοθέτημα αλλά η εφαρμογή του. Υπάρχει το θέμα της ευθυγράμμισης με τη Λισαβόνα βεβαίως Υπάρχει το ζήτημα ανάμεσα στο τι επιλέγουμε κατεχώρηση ή εκτελεστικές ε, πράξεις. Πάντως πρέπει να είμαστε σαφείς. Η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι η ευθυγράμμιση του ισχύοντος κανονισμού με την Λισαβόνα. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να ε, ε, συζητήσουμε και για την ίδια την μεταρρύθμιση έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον ίδιο τον κανονισμό. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν ε, μπορεί να μας πει δύο λόγια, αν έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή ε, τις εργασίες για την αναθεώρηση της ε, νομοθεσίας. Μπορεί οι εργασίες αυτές να γίνουν εκ παραλίλου, δεν αντιτίθεται η μία στην άλλη. Και βεβαίως μπορούμε συζητώντας για το θέμα που μας απασχολεί, της ευθυγράμμισης δηλαδή, να συζητήσουμε και ζητήματα που άπτονται της ε, μεταρρύθμισης. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ένα πρόβλημα υλοποίηση. Μερικές φορές είναι δημοσιονομικό το ζήτημα, άλλες φορές όμως είναι καθαρά ε, ε, θέμα το οποίο απορρέει από την διοικητική αδυναμία. Η συζήτηση του ΤΙΔΟ θα μας δώσει και τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε ε, κάποια άλλα θέματα. Ε, βέβαια τώρα μόλις διάβασα εγώ την, ε, ε, αυτό το προσχέδιο της έκθεσης, πρέπει να το μελετήσουμε, να το συζητήσουμε μεταξύ μας, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την τοποθέτηση της εισηγήτριας. Ευχαριστώ Ραούλ. Η Κάρμεν Φράγα έχει το λόγο. Ευχαριστώ την εισηγητρία. Η δουλειά της είναι δύσκολη. Κοιτούσα τον κανονισμό με τους βοηθούς μου στο γραφείο. Είναι πραγματικά πολύ περίπλοκος. Γιατί ε, τα όρια δεν είναι σαφή πάντοτε. Πολύ δε περισσότερο. Όταν ακούει κανείς ε, ε, τη συζητή στο Συμβούλιο. Είναι πολιτικά ευαίσθητα, πολιτικώς ευαίσθητα τα θέματα. Ακόμα και όταν δεν μπαίνουμε στην επιτροπολογία και πρόκειται για την ε, νομοθετική διαδικασία. Οπότε σε μικρέ ομάδε θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Δεν προτείνω να ασχοληθούν όλοι γιατί θα είναι πολύ βαρετό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση προ την Επιτροπή. Υπάρχει και άλλο κανονισμό, ο ο 404 νομίζω ε, που εξειδικεύει αυτόν τον κανονισμό. Πρόκειται για αυτό το δεύτερο κανονισμό, αυτός ο δεύτερος κανονισμός πρόκειται για ένα κανονισμό που είναι επιτροπολογίας. Οπότε ε, τι επιπτώσεις θα έχει η απόφαση που θα πάρουμε για την προσαρμογή στη Λισαβόνα στον άλλο κανονισμό που είναι 100% επιτροπολογία. Μπορεί να μην έχει καμία. Ας μου το εξηγήσει όμως η Κομισιόν. Τι θα γίνει με τον κανονισμό 404 γιατί εμπίπτει στην επιτροπολογία. Ε, θέλει κάποιος άλλος το λόγο, όχι, επομένως θα δώσω αμέσως τον λόγο στον Ενέστο Πάνια που εκπροσωπεί την Κομισιόν. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Τομά για αυτό το έγγραφο για μας είναι μια εξαιρετική βάση προκειμένου να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Το Σεπτέμβρη θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Είναι ο πιο περίπλοκος κανονισμός σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σε πώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, πολλή προσπάθεια και χωρίς να γνωρούμε το πόσο πολιτικά ευαίσθητο είναι το θέμα. Η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχουν σαφείς ε, περιπτώσεις, για παράδειγμα άρθρου 190 ή άρθρου 291. Τώρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει και μια φαιά ζώνη, μια γκρίζα ζώνη με μεγαλύτερο περιθώριο ερμηνείας. Εμείς από πού ξεκινάμε. Ε, θα πρέπει να βασιστούμε στη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του άρθρου 290 και του άρθρου 291 της συνθήκης. Ε, ερμηνείες του τύπου ε, ότι οι, ε, οι εκτελεστικές πράξεις εφαρμόζονται ε, για πιο τεχνικά θέματα και λιγότερο πολιτικά ε, η πράξη καταξιοδότηση για πιο πολιτικά θέματα, ε, μια τέτοια ερμηνεία θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλήξει αδιέξοδο στο Συμβούλιο. Ε, Ενδεχομένω δεν θα βοηθούσε μια τέτοια προσέγγιση σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικό τριμερή διάλογο. Για μας είναι πολύ σημαντική πολύ σημαντικό το δόγμα που έχει δημιουργήσει το Memorandum Συνεργασίας το μεταξύ των τριών οργάνων για την ερμηνεία των άρθρων 290 και 291. Κατά την άποψη της Κομισιόν όσο πιο πολύ μένουμε προσιλωμένοι σε αυτή την ε, διοργανική συμφωνία, τόσο πιο απλός και εύκολος θα είναι ο μελλοντικό τερμερής διάλογος. Ας το θυμόμαστε γιατί τα περιθώρια ερμηνείας έχουν πλέον περιοριστεί μέσω της διοργανικής αυτής συμφωνίας. Η κυρία Τομάς αναφέρεται στο θέμα της εναρμόνισης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό Συμμεριζόμαστε απολύτως το στόχο της ηγήτριας, αλλά να σας κάνω δύο παρατηρήσεις, μικρές επιφυλάξεις. Ε, πρώτον, υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί εναρμόνισης. δεν συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα την ίδια μικροδιαχείριση για όλες τις περιπτώσεις και για όλες τις περιοχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα υιοθέτησε μια πραγματικά σημαντική μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής με ένα καινούριο άξονα που είναι η περιφερειοποίηση. Συνεπώς όταν μιλάμε για εναρμόνιση θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μια εναρμόνιση απαιτήσεων προδιαγραφών προτύπων και εκεί συμφωνούμε αλλά ταυτόχρονα θα σας καλούσα να έχετε στο μυαλό σας ότι θα ξεκινήσουμε και μια διαδικασία περιφερειοποίησης. Οπότε η περιφερειοποίηση θα πρέπει να έχει ένα πραγματικό περιεχόμενο. Δεν θα πρέπει να είναι κοινή περιεχομένου. Αν οι κανόνες είναι τόσο ε, λεπτομερείς ε, κανόνες μικροδιαχείρισης θα είναι σαν να αφαιρούμε την ουσία από την περιφερειοποίηση. Ας βρούμε μια ισορροπία. Δεν είναι εύκολη η ισορροπία αυτή. Θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί προκειμένου η τροποποίηση αυτού τον κανονισμό ελέγχου να σεβαστούν το στόχο για κανόνες που θα είναι ισοδύναμη για όλους τους αλληλείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην δημιουργούνται δηλαδή διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα θα αφήνουν αυτοί οι κανόνες ένα αρκετό περιθώριο έτσι ώστε η περιφερειοποίηση την οποία θα ξεκινήσουμε να έχει περιεχόμενο, να έχει ουσία. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, και εδώ συμφωνούμε, με το στόχο της ε, κυρίας Από την άλλη μεριά, διαφάνεια ναι, αλλά η Κομισιόν, όπως θα θυμάστε, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για την μεταρρύθμιση, υποστήριξε όλες τις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αύξηση της διαφάνειας. Αποδείξαμε ότι είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ αυτού του στόχου, αλλά λίγο προσοχή με ορισμένα θέματα όπως για παράδειγμα την ιδέα ε, διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, μέτρα τα οποία ε, θα ε, αλλοιώνουν τι αρμοδιότητε μα και τα καθήκοντά μα σύμφωνα με τι συνθήκε. Ε, οι υποχρεώσει της Κομισιόν θα πρέπει να αυτέ που προβλέπονται από τη συνθήκη στο πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων και των πράξεων κατά Τώρα, παρόλο ότι δεν υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους μας, ε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στόχο τη Κομισιόν είναι σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στα θέματα ελέγχου, ε, η Κομισιόν, λέω, είναι αποφασισμένη να διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους. Χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό βέβαια για μας. Και εκεί μπαίνουν και τα ΡΑΚ. Για μας είναι επίσημα σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε στην, στο, στόχο για τον οποίο γίνεται αυτή η δουλειά. Δηλαδή ο στόχος δεν είναι να αμφισβητηθούν οι, οι κανόνες ελέγχου που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Που έτσι κι αλλιώς είναι καινούργοι. Ε, ο στόχος είναι να προσαρμοστεί ο κανονισμός της συνθήκη της Αβώνας. Οπότε δεν θα ήταν σκόπιμο, πιστεύει η Κομισιόν, να επωφεληθούμε τη συζήτηση για να ε, υιοθετήσουμε προτάσεις που δεν έχουν σχέση με τον έλεγχο. Προτάσεις ενδεχομένω εύλογε, λογικές, χρήσιμες κλπ. Αλλά που δεν έχουν σχέση και δεν εμπίπτουν στην ευθυγράμμιση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γιατί αν στην περιπλοκότητα του κανονισμού προσθέσουμε την πρόσθετη περιπλοκότητα προτάσεων οι οποίε δεν έχουν σχέση με την προσαρμογή στην θήκη της Λισαβόνα, ε, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ αργότερα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για θέματα όπως η ασφάλεια στα λιευτικά σκάφη, μην ξεχνάμε ότι πέραν της περιπλοκότητας που προσθέτουμε, δημιουργούνται και νομικής φύσεως θέματα. Ας περιοριστούμε λοιπόν στην λησβονοποίηση του κανονισμού. Τώρα για τις ερωτήσεις Ρωμέβα και Φράγα. Για την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Ε, έτσι κι αλλιώς ο κανονισμός αυτός είναι πρόσφατος. Αυτή τη στιγμή τον εφαρμόζουμε, βρισκόμαστε σε δικασία εφαρμογής του. Μην ξεχνάτε ότι ορισμένες διατάξεις δεν ετέθησαν σε εφαρμογή αμέσως μετά την ε, υιοθέτηση του κανονισμού. Είχαμε μια ε, μεταβατική περίοδο ενός ή δύο ετών, ε, οπότε αυτή τη στιγμή η δυο ετων οποτε αυτη τη στιγμη η τροποποιηση του κανονισμού δεν βρίσκεται στα σχέδιά μας. Θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε και μετά να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Φράγα. Όλη αυτή η διαδικασία θα έχει την εξή συνέπεια. Ο κανονισμός αυτός, ο εφαρμοστικός κανονισμός, α, αν ε, ο αριθμός των τροποποίησεων του κανονισμού βάσης είναι σημαντικός, και καταστήσει απαραίτητη την τροποποίηση του εφαρμοστικού κανονισμού, τότε η Κομισιόν θα αναθεωρήσει τον εφαρμοστικό κανονισμό με, μέσω, με δύο κανονισμούς. Δηλαδή θα τον χωρίσουμε σε δύο τμήματα, ένα κανονισμό με τις κατεξιδότητες πράξεις και ένα κανονισμό με τις ε, ε, εφαρμοστικές πράξεις. Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση θα ήθελα μονάχα, αγαπητέ Έρνεστο. Έχει μας εμπιστοσύνη, εμείς θα φτάσουμε την ευθυγράμμιση με τη Λισαβόνα μέχρι τέλους, μέχρι τελευταίας ρανίδας. Μην έχει καμία αμφιβολία. Θα δώσω το λόγο ξανά στην Ιζαμπέλ Τομά, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η εντελεγή απόψεων στα έγγραφο εργασία τη η κυρία Τόμα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για την συνεισφορά τους ε, και για να απαντήσω στην πρόταση της κυρίας Φράγα ε, να πω ότι όντως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια συνάντηση εργασία τον Σεπτέμβρη με τους σκιώδεις για όσους βεβαίως είναι πρόθυμοι να ε, ε, κάνουν την εργασία αυτή πριν σταλεί στην μετάφραση η έκθεση έτσι ώστε να έχουμε ε, όσο γίνεται περισσότερο συνεργαστεί μεταξύ μας. Δεύτερον, για να απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Πένια Διάδο. σχετικά με το ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε την ευθυγράμμιση με τη Λισαβόνα. Αλλά παρόλα αυτά να πω ότι ο ρόλος που έχουμε σε, αυτήν την, σε αυτόν τον ρόλο ε, ε, καθορισμού ε, της διαδικασίας της υλοποίησης των μέτρων ελέγχου. Ο ρόλος, λέω, είναι πολιτικός πρωτίστως και οπωσδήποτε στις κατεξουσιοδότηση πράξεις έχουμε την ευθύνη να ε, προσανατολίσουμε την Κομισιόν, μια και έχουμε υποχρέωση ελέγχου εκ των υστέρων. Άρα εκ των προτέρων προσανατολίσουμε την Κομισιόν για τους εκ των υστέρων ελέγχους που θα κάνουμε. Είναι σωστό, είναι ορθό να ε, οδηγήσουμε την Κομισιόν, να την προσανατολίσουμε ε, στην καλύτερη οδό. Και είναι σωστό αυτό που είπε ο συνάδελφος Ραούλ προηγουμένως. γιατί αυτός είναι ο κύριος άξονας ε, της ευθυγράμμισης με τη Λισαβόνα. Επίσης, σε σχέση με την περιφερειοποίηση, ε, που είναι ιδιαίτερος προσφυλής, όπως ξέρετε αγαπητέ κύριε Πενιαζιάδο, η συνεργασία ε, με τα περιφερειακά συμβούλια που είναι και πρόταση που κάνω όσον αφορά τις της πράξεις άλλωστε πιστεύω το εξής πρώτον ο προσανατολισμός του Κοινοβουλίου ε, που μπορεί να δώσει δηλαδή το Κοινοβούλιο στην Κομισιόν μπορεί να περιλαμβάνει και αυτήν την σύσταση έτσι ώστε η απόφαση για κατεξουσιοδότηση πράξη να εγκριθεί από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και δεύτερον πάντως αναφορά την περιφερειοποίηση ή μάλλον την μικροδιαχείριση, γιατί αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιήσατε. Εκεί, αντιθέτως, πιστεύω ότι όσον αφορά τον έλεγχο, και το τονίζω, όσον αφορά τον έλεγχο, δεν θα ήταν καλό, κατά την άποψή μου, να ε, ε, δούμε έτσι διαφορετικά ειδικούς ε, ε, ρόλους ή τρόπους ε, για, τα, για τις θαλάσσιες λεκάνες. Γιατί επαναλαμβάνω η δυσπιστία και των επαγγελματιών του κλάδου και των πολιτών με τον τρόπο αυτό θα ενισχύεται. Υπάρχει διαφορά προσέγγισης και στις εκτελεστικές ε, ε, πράξεις οπωσδήποτε θα υπάρξουν ιδιαιτερότητες φυσικά, αλλά ε, όσον αφορά το μεγαλύτερο μέρος του, του ελέγχου νομίζω ότι δεν θα πρέπει να προωθήσουμε τις ιδιαιτερότητες. Αντιθέτως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ομοιογένεια έτσι ώστε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και του κλάδου. Ευχαριστώ. Ε, παρουσίαση της έκθεσης 15 Οκτωβρίου. Μετά την, ε, ε, και μετά η διαδικασία θα συνεχιστεί. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα αλλάξουμε ε, ομιλήτρια. Θα μιλήσουμε τώρα για τον προγραμματισμό του, του θαλάσσιου χώρου και ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτήων ζωνών με εισηγήτρια πάντα την κυρία Ιζαμπέλ Τομάς. Προτείνω ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος αυτού. Σου δίνω το λόγο Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Όντω. Εδώ έχουμε σχέδιο οδηγίας που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μετά τις δηλώσεις της ε, Λευκοσίας ε, και διαστόματος των αρμοδίων υπουργών ε, απεφάσισε ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στα πλαίσια της ε, γαλάζιας ανάπτυξης και της στρατηγικής 2020 επικυρώνοντας την απόφαση για υλοποίηση αυτής της γαλάζιας ανάπτυξης. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση της γαλάζιας ανάπτυξης. Άλλωστε τα συζητήσαμε αυτά και με την έκθεση πρωτοβουλίας κυρίας Πατράου Νάβες λίγο πιο ε, νωρίς ε, σήμερα. Η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η περιπλοκότητα των ε, χρήσεων μπορεί δυστυχώς συχνά να οδηγήσει σε ε, εμπλοκές και παρεμποδίσεις της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων. Όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχουν οι παλαιές βλέπε ε, ε, από χιλιετιών παραδοσιακές χρήσεις, αλλά υπάρχουν και νέες δραστηριότητες οι οποίες προστίθενται Βεβαίως αναφέρομαι και στην θαλάσσια ενέργεια, αλλά ενδεχομένως και οι εξορίξεις διαφόρων ειδών και τα λοιπά, ή ε, η χρήση των ΑΟΖ και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς ε, μπορούμε να συνεχίσουμε ε, την ε, ε, χρήση χωρίς όμως να υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων, συγκρούσεις όσον αφορά την διατήρηση των θαλασσών, όσον αφορά την ανάπτυξη και πώς όλες αυτές οι διενέξεις είτε να αποφευθούν είτε να μπορούν να επιληθούν με ένομα μέσα. Έχουμε πρόταση της Κομισιόν που ζητά ε, από τα κράτη-μέλη να ε, προχωρήσουν σε ε, χωροταξία του θαλάσσιου χώρου, καθώς επίσης και ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτήων ζωνών, ε, δηλαδή από τη μία πλευρά δεν υπάρχει πλέον κατάτμιση των ζωνών επιτρέποντας ε, διάφορες παραχωρήσεις ε, χωρίς να ληφθεί υπόψη η χρήση των άλλων. Από την άλλη πλευρά αναφερόμαστε σε ολοκληρωμένες θαλάσσιες πρακτικές και ταυτοχρόνως θέλουμε και μία διακυβέρνηση η οποία θα επιτρέπει την διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η πρόταση οδηγίας ε, της ε, Κομισιόν βασίζεται σε υφιστάμενες οδηγίες, ε, κυρίως αυτό, αυτή είναι της στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο και άλλες οδηγίες που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς επίσης και τα σχετικά με την ενεργειακή ανάπτυξη και μπορεί να ληφθεί ληφθεί, να ληφθούν όλα τα στοιχεία αυτά ως νομική βάση για αυτό το σχέδιο οδηγίας. Τι άλλο να σας πω. Α, έχω ξαναπεί στην Επιτροπή Αλληλείας ότι είμαι πεπισμένη ότι αν θέλουμε να δούμε μια πραγματική ανάδυση της γαλάζιας ανάπτυξης και αν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε στη δημιουργία του 1,5 εκατομμυρίου επιπλέον θέσεων εργασίας ε, ε, μέχρι το 2014 ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα χωροταξίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, έστω και αν, όπως είπαμε και σήμερα το πρωί, πρέπει να διαθέτουμε συγκεκριμένα και σωστά δεδομένα για να το επιτύχουμε. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά και κυρίως μια και το ζήτημα έχει τεθεί πλέον, δηλαδή του να ε, ξέρουμε εάν η οδηγία είναι το κατάλληλο μέσο. Μπορώ να πω ότι κυρίως όσον αφορά το θαλάσσιο χώρο ε, ε, έχουμε ζώνες οι οποίες στις οποίες μάλλον ασκούνται διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες μάλιστα ασκούν διαφορετικά κράτη-μέλη και επομένως η ιδέα του χώρου είναι τέτοια που εάν δεν έχουμε είτε όμοια εργαλεία είτε συναφή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα της θαλάσσης ε, διακρατικά θα έχουμε πρόβλημα. Επομένως η εναρμόνιση είναι κάτι θετικό. Επίσης, θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη-μέλη, αν πραγματικά θέλουν τη γαλάζια ανάπτυξη, θα πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα και έστω και αν η χωροταξία και η ολοκληρωμένη διαχείριση πρέπει να αφήνει σημαντικό περιθώριο και στις ε, χώρες ε, μέλη, γιατί πολλές ε, ε, από τις χώρες έχουν ε, ήδη προχωρήσει σε ολοκληρωμένη διαχείριση ή χωροταξία ε, του θαλάσσιου χώρου, επομένως δεν χρειάζεται να ξαναρχίσουν τη δουλειά τους από το μηδέν. Επίσης γνωρίζουμε ότι κάποιες, άλλες χώρες, κάποιες χώρες έχουν ε, κεντρική διακυβέρνηση, άλλες πιο περιφερειακή και αποκεντρωμένη. Ε, θα πρέπει να σεβαστούμε βεβαίως και τα θεσμικά όργανα της κάθε χώρας. Από την άλλη πλευρά και αυτό σίγουρα θα ε, ε, αποτελέσει και αντικείμενο τροπολογίας που θα υποβάλω στην Κομισιόν, στο κείμενο της Κομισιόν. Οι εμπλεκόμενοι είτε είναι τοπικές και περιφερειακές αρχές, είτε είναι οι εργαζόμενοι επαγγελματίες του κλάδου, λοιπόν λέω όλων των ε, ε, εμπλεκομένων φορέων είναι εκ των ουκάνε προϋπόθεση για το σωστό προγραμματισμό του θαλάσσιου χώρου και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Είναι απαραίτητα μέρη της ε, υλοποίησης των προαναφερθέντων. Τελευταία παρατήρηση προς την Κομισιόν. ο κατάλογος των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να βάλουν τα κράτη-μέλη στον προγραμματισμό και το χωροταξία του θαλασσίου χώρου. Ξέρω ότι μέχρι τώρα υπάρχει περιορισμός στις θαλαμοδιότητες της ε, Ένωσης, αλλά εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, οπωσδήποτε θα πρέπει να βάλουμε και την αναψυχή και τον τουρισμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε ε, και την ε, μεταλλευτική εξόριξη. γιατί διαφορετικά εάν ασχοληθούμε μονάχα με κάποιες χρήσεις και όχι με όλες, τελικά δεν θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε τις συγκρούσεις ε, που απορρέουν από τις διαφορετικές χρήσεις. Βεβαίω έχουμε τι ανοσιακέ αρμοδιότητε, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε μια εξαιρετικά περιοριστική λίστα, η οποία δεν θα επιτρέψει την επίλυση των προβλημάτων τελικά. η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι και επομένως θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά και όλες τις χρήσεις στην χωροταξία του θαλάσσιου χώρου και την ολοκληρωμένη διαχείρισή του. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, υπενθυμίζω ότι πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας ε, και ε, η Επιτροπή Μεταφορών είναι η αρμόδια επί της ουσίας. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Κοσλόφσκι, ο οποίος ε, ζήτησε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του κυρίου Βαλέσα θα λάβω το λόγο που είναι απόν. Θα διαβάσω την δήλωσή του η ανάπτυξη και εντατικοποίηση της ανθρώπινης δραστηριότητα στη θάλασσα συμβάλλει ε, στην αναδιοργάνωση του χωροτοξικού, χωροτοξικού σχεδιασμού ε, και ε, δημιουργεί νέες ισορροπίες και ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα κράτη-μέλη ε, έχουν αρχίσει στον παράκτιο χώρο να καταρτίζουν προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών τους τα κράτη-μέλη έχουν σύντομη προθεσμία για την κατάρτιση ε, εγγράφων. Χρειάζεται επίσης να υποβάλουν εκθέσεις και αυτό δημιουργεί σε εθνικό επίπεδο δυσκολίες στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων. Δηλαδή ε, είναι πρόσθετος ο φόρτος στα κράτη-μέλη. Ο επιχειρησιακός στόχος ε, υλοποιείται από τα έγγραφα αυτά αλλά δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία ε, συχνά από αυτό το εγχείρημα. Θα πρέπει να ε, υποστηρίξουμε την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια. Αυτός ο στόχος στα πλαίσια της ε, κοινής αλληλευτικής πολιτικής ε, προωθείται και έγιναν μετά την τελευταία μεταρρύθμιση πολλές εντατικές εργασίες. Πολλά εθνικά κοινοβούλια και το πολωνικό ε, θεωρούν ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα με την επικουρικότητα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει με βάση τις τομεακές πολιτικές ε, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αλίας ε, να μην ε, προβλέπονται επιδοτήσεις οι οποίες δεν θα κρυθούν σκόπιμες. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ Βενζιδί, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ιζαμπέλ Τομά για την εξαιρετική εισαγωγή στο θέμα. Γιατί χρειάζονται δηλαδή ε, τα μέτρα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γι' αυτό ε, είναι ενδιαφέρουσα η κοινή πολιτική αλίας, γιατί μας, μας απαιτεί να γίνουμε πιο ρεαλιστές και να συνεργαζόμεθα. Ο συνάδελφος από την Πολωνία είπε ότι πολλά κράτη-μέλη φαίνεται να έχουν προβλήματα με την προτινόμενη αυτή οδηγία, γιατί παρεμβαίνει σε αυτό που θεωρούν προνόμια των κρατών μελών. Ε, και εδώ έχουμε μια πρόκληση να αντιμετωπίσουμε στη θαλάσσια πολιτική. Βεβαίως, ε, οι χερσαίες δραστηριότητες σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν και τη θάλασσα και αν θέλουμε επιτυχή θαλάσσια πολιτική και βεβαίως δεν είναι μόνο η Βαλτική που έχει περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και η Μεσόγειος και ο Ατλαντικός λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε τις θάλασσές μας που δεν είναι υγιείς τι θα κάνουμε αν κάνουμε κάτι θα επηρεαστεί η πολιτική γεωργία. Μια σειρά πολιτικών θα επηρεαστούν που λαμβάνουν χώρα στην ξηρά. Και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση προφανώς γιατί για να γίνει κάτι για τη θάλασσα πρέπει να κοιτάξουμε και την ξηρά. Και ο θαλάσσιος σχεδιασμός σημαίνει μεταξύ άλλων ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε περισσότερο παράκτιο σχεδιασμό. Είναι ε, λεπτό λοιπόν το θέμα για πολλές χώρες μέλη και για τη δική μου τη Σουηδία που έχει πάρει θέση πάνω σε αυτό το θέμα και πιστεύει ότι πραγματικά υπησέρχεται πολύ το θέμα αυτό στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό είναι κρίμα όμως γιατί Χρειαζόμαστε κοινή υποβολή εκθέσεων, εναρμόνιση ε, στη συλλογή των δεδομένων. Πρέπει να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, γνωμοδοτήσεων, γιατί είμαστε γείτονες και πρέπει να προσεγγίσουμε από κοινού το θέμα. Στη Βαλτική το βλέπουμε. Δεν γίνεται τίποτε αν η Σουηδία δραμώνει δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και με τη Ρωσία θα πρέπει να γίνουν κοινές προσεγγίσεις, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται στη Βαλτική. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Ενώ και κά... κάποιες χώρες θεωρούν ότι η δουλειά γίνεται. Η Σουηδία όμως δεν έχει καν αρχίσει τον ε, θαλάσσιο σχεδιασμό. Οπότε δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με βάση την οδηγία. Εγώ προβλέπω ότι το θέμα θα είναι ε, αμφιλεγόμενο σε σχέση και με την οδηγία για το θαλάσσιο σχεδιασμό και θα υπάρξουν χώρες μέλη που θα θεωρήσουν ότι η οδηγία επισέρχεται στα δικά τους δικαιώματα και αρμοδιότητες. Θα γίνει λοιπόν η συζήτηση, θα δούμε πού θα βάλουμε τα όρια και πού πρέπει να επιμείνουμε όπως ε, στις εκθέσεις, ε, στους στόχους ε, αυτά δεν πρέπει να είναι επίμαχα θέματα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιους κοινού στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για την ε, θαλάσσια στρατηγική. Όλα αυτά είναι κομμάτι της στρατηγικής 2020 και εδώ έχουμε τα μέσα για να επιτευχθούν οι στόχοι. Τώρα, μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά την πρόταση της Κομισιόν και που αφορά το άρθρο 8 όπου έχουμε κατάλογο θεμάτων που πρέπει να συμπεριληφθούν στο ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Έχουμε ανανεώσιμη ενέργεια, γεωργία, αλληλεία και άλλα. Αλλά ένας από τους σημαντικότερους τομείς που αφορά τις παράκτιες ζώνες είναι ο κλάδος του τουρισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της οικονομίας μας. Ο τουρισμός ε, περιλαμβάνει πολλούς τομείς. Και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό μας όπως τα λιμάνια και η εξέδραση εξόριξης. Γιατί λοιπόν δεν έχει συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ. Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Μεταφορών ασχολούμεθα άμεσα με το θέμα και είναι η συγγήτρια εκεί η συνάδελφος Μάη Συνεργιά το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ασχοληθήκαμε εντατικά με τους επιμέρους τομείς εκεί, δηλαδή η πολυλειτουργική χρήση των θαλασσών που αποτελούν μια ευρύτερη διάσταση και πιστεύουμε ότι πρέπει στη χρήση των πόρων να προχωρήσουμε με σύντονο τρόπο. Από την άλλη δεν θέλουμε πρόσθετο επίπεδο ευρωπαϊκού σχεδιασμού όπου όλες οι δραστηριότητες των κρατών μελών θα πρέπει να χρήζουν έγκριση προτέρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το παρουσιάζει η συνάδελφος Τωμά πολύ ωραία που λέει ότι χρειάζεται ελευθερία για τα κράτη-μέλη μας. Ε, περνάμε τώρα από δύσκολη οικονομική συγκυρία και οι δυνατότητες των θαλάσσιων πόρων για αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία απασχόλησης είναι τεράστιο. Τεράστιες δυνατότητες υπάρχουν εκεί. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχει ένα εθνικό επίπεδο το οποίο θα έχει καλό μηχανισμό σχεδιασμού και όπου θα συντονίζονται οι επιμέρους τομείς. Στην Αλία, για παράδειγμα, έχουμε τα 12 μίλια τη ζώνη προστασίας ελίας, τρία ναυτικά μίλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, σε οτιδήποτε είναι διασυνοριακό. Ε, μετά έχουμε τις ΑΟΖ, που ε, φτάνουν μέχρι τα διεθνή ύδατα και αν υπάρχουν ε, έργα διασυνοριακά θα πρέπει να συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, σε, επίπεδο ευρωπαϊκού σχεδιασμού νομίζω ότι συμφωνούμε εδώ και με, τον, ε, με τους συναδέλφους Κοσλόφσκι και Βαλέσα. Βέβαια υπάρχουν και διαφορετικοί τομείς όπου εκεί μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις. Έχουμε τις θαλάσσιες οδούς ναυσιπλοείας, αν δούμε δηλαδή τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, Βορεια Θάλασσα. Ε, ε υπάρχουν ε, προφανώς κάποιες προτεραιότητες εκεί, αλλά θα πρέπει να τηρούνται και οι περιβαλλοντικοί όροι προστασίας. Τώρα μπορεί να είναι Natura 2000, μπορεί να είναι περιοχές FFA, ε, άλλες σημαντικές προστατευόμενες περιοχές, όλα αυτά πρέπει να τηρούνται. Στις ε, ζώνες αλληλείας είναι πολύ σημαντικό να ορίζονται, να οριοθετούνται και εμείς ως Επιτροπή Αλληλείας καθήκον έχουμε να φροντίσουμε για την προστασία τους και να μην υπάρχει καμία σύγκρουση εκεί, γιατί αυτές θα είναι οριοθετημένες, έχουμε δηλαδή τις ε, ζώνες, τις προστατευόμενες των αποθεμάτων, ε, νεαρών ψαριών και κλπ. Ε, ζώνες αναπαραγωγής των ηχθείων. Ο τουριστικός τομέας οπωσδήποτε συνιστά σημαντικό οικονομικό παράγοντα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά εδώ ε, μιλάμε και για διασυνοριακά προγράμματα, ένα μεγάλο πρόγραμμα ας πούμε που εμπλέκει περισσότερα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, ε, βρίσκεται σε επίπεδο σχεδιασμού ευρωπαϊκού. Τέλος, να τονίσω ότι ορίζουμε διαδρόμους εδώ που θα υπάρχουν για μέτρα υποδομών. Ε, όταν πρόκειται για ηλεκτροδότηση, όταν πρόκειται για αγωγούς αερίου, ε, ε, για εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας. Όλα αυτά πρέπει να συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς θα, είναι, πώς θα κατασκευαστεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης, να μην έχουμε επίσης για νέα χάραξη πάντοτε τις παλιές μεθόδους αλλά να είμαστε πιο συντονισμένοι. Ε, νομίζω ότι και η κυρία Μάισνερ τα έχει λάβει υπόψη αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ που είναι η συγκεκριμένη. Ε, και επομένως, ε, μια και είναι και αρμόδια από την Επιτροπή Μεταφορών, να μας τα πει. Ευχαριστώ. Ναι, είμαι εδώ με διπλή ιδιότητα στην Επιτροπή Μεταφορών Εισηγήτρια, εδώ σκιώδης. Συγγνώμη Ιζαμπέλ που καθυστέρησα να έρθω και να ακούσω την ε, παρουσίαση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλίας. Ε, έχουν συζητηθεί όμως αυτά. Ε, είχα και άλλη μια υποχρέωση και καθυστέρησα λίγο παρόλο που ήλπιζα να προλάβω. Τα μετά τα άκουσα. Πράγματι, από τη σκοπιά της Επιτροπής Αλίας είναι σημαντικό κυρίως να δούμε τι ρόλο παίζει η Αλία στην ανάπτυξη ε, του θαλάσσιου χώρου, στην κατανομή και, τι, θα πρέπει να έχει τη θέση που της αξίζει. Βέβαια η Επιτροπή ενδιαφέρεται και για τη θάλασσα γενικότερα και αυτό είναι το αγαπημένο μου θέμα από τότε που ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 πολύ συνειδητά γιατί είδαν ότι όλο και περισσότερες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στη θάλασσα και στο βυθό των θαλασσών. Και η θάλασσα έχει μια οικολογική ζώνη πολύ ευαίσθητη και πρέπει να τη φροντίσουμε και για χάρη των νέων, των επομένων γενεών ε, θα πρέπει να φροντίσουμε για τη βιωσιμότητα, διατηρησιμότητα, η φορεία των θαλασσών, την υγεία των θαλασσών. Και αυτό συνεπάγεται προστασία ευαίσθητων ζωνών. Ε, σε ορισμένε περιοχέ τα καταφέραμε. Εγώ είμαι από την κάτω Σαξονία, στο Βάτενμερ στη Γερμανία, που είναι μια μοναδική ζώνη προστατευόμενη και υπάρχει εκεί βιώσιμο τουρισμό και τους εξηγούμε την αξία της θάλασσα και του οικοσυστήματος. Ε, ε, βεβαίως υπάρχει αλληλεία, υπάρχει ναυσιπλοεία και ε, στις ακτές των νησιών υπάρχουν και εξέδρες εξόρισης. Όλα υπάρχουν, δεν αναποκλείεται τίποτα και λειτουργούν όλα πολύ καλά και ρυθμίζονται ε, με τρόπο συντονισμένο, ε, με συμφωνίες, υπήρξαν πολλές συμφωνίες με, με πολλούς φορείς. Είναι λοιπόν λογική απόρρια από την, της ολοκληρωμένης πολιτικής της θάλασσας ότι όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούμε τα μέσα αυτά. Από την αρχή του 2007 ήδη συζητούσαμε για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Αυτό το συμφώνησαν από την αρχή όλα τα κράτη-μέλη. Και τώρα έχουμε και την πράσινη ανάπτυξη, είχαμε το ENP, που είναι η θαλάσσιο, ο θαλάσσιος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 που θέλουμε να φροντίσουμε για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτά που υπάρχουν λοιπόν και αυτό προσπαθεί να κάνει η Κομισιόν στην πρότασή της. Αυτά που υπάρχουν σε σχέση με θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και διαχείριση παράκτιων ε, ζωνών και προστασία των ευαίσθητων ζωτών, ζωνών, πώς μπορούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε σε μια πιο χαλαρή, όπως είπε η Κομισιόν, οδηγία πλαίσιο. Σε μια άλλη συνάντηση το είχε πει αυτό. Βεβαίως ε, καταλαβαίνουμε τα κράτη-μέλη που μπορεί να πούν δεν θα μας υπαγορεύει η Ευρώπη τι θα κάνουμε εμείς. Μπορούμε και μόνοι μας, το λέω έτσι τώρα λίγο ε, πρόχειρα. Αλλά παράλληλα η Κομισιόν ήδη στον πρόλογο της γράφει ότι δεν θέλει να υπαγορεύει πολλά πράγματα αυτά που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν, θέλει να τα αξιοποιήσει. Και στην έκθεσή μου που τη συντάσω τώρα και θα πάει αύριο να μεταφραστεί, έχω προχωρήσει πολύ, και ε, έκανα ανταλλαγέ απόψεων με πολλού συναδέλφου. Θα αποσαφηνίσω κάποια πράγματα γιατί δεν είναι αλήθεια ότι ε, ε, η Κομισιόν γράφει ότι όλα αυτά που υφίστανται δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε και δεν θέλουμε να φτιάξουμε νέε γραφειοκρατίε, νέε στρατηγικέ. Ε, όταν τα κράτη-μέλη ήδη έχουν υφιστάμενα προγράμματα και σχέδια διαχείρισης κλπ. Δεν θέλουμε πρόσθετα. Καμιά φορά δεν φαίνεται αυτό από το άρθρα της πρότασης. Πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό. Τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε όλα τα παράκτια κράτη στην Ευρώπη, όσοι έχουν να κάνουν με παράκτιες ζώνες, γιατί υπάρχουν κράτη που δεν έχουν ε, ακτές, αλλά με κάποιο τρόπο συνδέονται με παράκτιες δραστηριότητες. Όλοι τέλο πάντων θα πρέπει να κατακτήσουν σχέδια και θα να δουν πώς μπορούν με τον καλύτερο τρόπο ε, να συμμετέχουν και να αποφύγουν ε, συγκρούσεις στο μέλλον και να φροντίσουν τα οικοσυστήματα. Υπάρχουν και άλλα συστήματα όπως κοινή διακυβέρνηση διασυνοριακή συνεργασία βεβαίως και όπως είπατε και συνεργασία με τρίτες χώρες. Δυστυχώς δεν άκουσα όπως σας είπα αυτά που είπε η Ζαμπέλ, αλλά μπορώ να τα φανταστώ τι είπε γιατί είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ μας και περιμένω με χαρά τη συνέχιση των εργασιών πάνω στην έκθεση αυτή και θα περιμένω με ενδιαφέρον και τις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Θα συνεχίσω να εργάζομαι πάνω σε αυτό το θέμα στην Επιτροπή ακόμα και όταν τελειώσουμε με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. <laughs> Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και στην ε, εισηγήτρια για αυτή την θετική και επικοδομητική εισαγωγή και για τη, την πολύ καλή συζήτηση. Έχω την εντύπωση πως ε, επικρατεί ένας κοινό φόβος. Να διευκρινίσω λοιπόν ορισμένα συστήματα. Ε, σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των δραστηριοτήτων και των τομέων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 8 της πρότασης. Να διευκρινίσω το εξής. Ο κατάλογος, οι που εμφανίζουν σε, αυτούς τους δύο, σε αυτά τα δύο άρθρα δεν είναι ε, εξαντλητικοί. Δεν αποκλείεται τα κράτη-μέλη να εισάγουν και ε, άλλες πολιτικές ε, που επιθυμούν. Εμείς μπορούμε να περιλάβουμε μόνο τους τομείς ε, στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα. Αλλά ο, η ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Αν για παράδειγμα θεωρείτε ότι ο τουρισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις παράκτητες περιοχές της, μπορεί να το συμπεριλάβει όπως και οποιοδήποτε άλλο τομέα. Τα κράτη-μέλη διατηρούν πλήρη αρμοδιότητα για το τι και πού θα προγραμματίσουν, ε, θα σχεδιάσουν χωροταξικά. Εμείς κατονομάσαμε αυτούς τους ε, τομείς ε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικοί με βάση τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δεν προκύπτουν νέες ε, τομεακές υποχρεώσεις, όχι, ήδη υπάρχουν οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες για αυτούς τους τομείς και γι' αυτό τους συμπεριλάβαμε. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη έχουν ένα περιθώριο λιγμών αρκετά πλατή. ο προγραμματισμός θα παραμείνει, ο σχεδιασμός θα παραμείνει ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Κομισιόν δεν πρόκειται να παρέμβει ούτε στον σχεδιασμό ούτε στη στρατηγική ούτε στη στρατηγική της διαχείρισης των παράκτιων ζώνων. Αυτά που εμείς έχουμε εδώ κατονομάσει, απαριθμίσει, είναι οι διαδικαστικής φύσεως υποχρεώσεις, έτσι ώστε ο σχεδιασμός να γίνει με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, με βάση συγκεκριμένους παράγοντες, κριτήρια και μέσω διασυνορική συνεργασία, διότι πολλέ από αυτέ τι δραστηριότητε απαιτούν τη διασυνοριακή συνεργασία. Πρόκειται για διαδικαστικές διοικητικές υποχρεώσεις, όχι υποχρεώσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του σχεδιασμού, την ουσία του. Σε ό,τι αφορά την κυρία Μέσνερ τώρα. Θα επαναλάβω ότι η οδηγία δεν απαιτεί από τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τις, ε, τη δομή της τοπικής ή κυβέρνησης ή και εθνικής κυβέρνησης. Τα κράτη-μέλη θα καθορίσουν μία περισσότερες αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνε για τη συνεργασία, θα έρχονται σε επαφή με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών, μελών ή τρίτων χωρών, αλλά και λέμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί καινούργιο επίπεδο διοίκησης. Θέλουμε να σεβαστούμε όλα όσα υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη, όλους τους μηχανισμούς, την, τους μηχανισμούς περιφερειακής και άλλους μηχανισμούς που ήδη υφίστανται. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε ένα ακόμα επίπεδο ε, γραφειοκρατίας ε, ή να απαιτήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή όταν ήδη υπάρχουν μηχανισμοί. Γιατί υπάρχουν και κράτη-μέλη στα οποία δεν υφίστανται τέτοιοι μηχανισμοί, οπότε θα υποχρεωθούν να ξεκινήσουν ε, να στήσουν μια διαδικασία διαβούλευσης, να ορίσουν αρμόδιες αρχές κλπ. Αλλά εκεί που ήδη υφίστανται τέτοιου είδους μηχανισμοί, τέτοιου είδους συστήματα, η πρότασή μας δεν πρόκειται να επιφέρει καμία αλλαγή, δεν πρόκειται να προσθέσει καμία υποχρέωση ή γραφειοκρατική ε, διαδικασία. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην Ιζαμπέλ Τομά για να ολοκληρώσει την παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα να καθησυχάσω τον κύριο Κοσλόφσκι και ε, μάλλον δια του κύριου Κοσλόφσκι τον κύριο Βαλέσα. Φρονώ ε, κυρίως ότι ο στόχος είναι εν τέλει επένδυση για την ανάπτυξη. Και όχι ένα επιπλέον κόστος ε, απλώς γιατί κάνουμε κέφι να, προγραμμα... να, χωροτα... να κάνουμε τη χωροταξία του... και το σχεδιασμό του θαλασσίου χώρου και ολοκληρωμένες διαχειρήσεις κτλ. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί, πολλά παραδείγματα στη χώρα μου, ακριβώς γιατί δεν είχε υπάρξει προγραμματισμός της χωροταξίας και δεν είχαν προβληθεί μελλοντικέ ε, χρήσεις ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο εκ των υστέρων να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Και να πω και στον κύριο Κούνο ότι συμφωνώ απολύτως συμφίνε κάθε χώρα μέλος θα πάρει τι αποφάσεις της και άλλωστε αυτό ε, λέει και επαναλαμβάνει και η Κομισιόν. Απλώς η οδηγία δεν ε, θα πρέπει να υποχρεώνει παρά μονάχα ε, το, τη διαδικασία προγραμματισμού και χωροταξίας, δηλαδή όχι τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Ε, δεν μπορεί να πει η οδηγία ποιες θα είναι οι ζώνες οι οποίες θα είναι ζώνες προστατευόμενες ή ποια δραστηριότητα θα λάβει χώρα που κτλ. Αυτά δεν είναι αρμοδιότητες της Ένωσης. Αντιθέτως, και ακριβώς εκεί έγκυται και η δυσκολία του εγχειρήματο, εάν ο καθορισμός της ε, χωροταξίας είναι επιβεβλισμένος και συμφωνώ ε, ε, με αυτά που λέει η κυρία Λέβιν για το άρθρο 5 γιατί κυρίως λέμε πρέπει να ασχοληθούμε με την αλληλεία εδώ, είναι σαφές ότι οι αλληλείς ενδιαφέρονται, είναι αυτοί που περισσότερο τους ενδιαφέρει η, η, όποια νέα δραστηριότητα στη θάλασσα και ο αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα είτε στις παράκτιες είτε περιοζώνες είτε και λίγο πιο ανοιχτά ας πούμε εξόριξη ή ε, λιμένας αναψυχής, ε, όλα αυτά ε, βεβαίως έχουν άμεσο και μεγάλο αντίκτυπο στους αλλιευτικούς πόρους και για να μην αναφερθώ στα ειδικά προβλήματα της θαλάσσιας ενέργειας και των πεδίων θαλάσσιας ενέργειας κτλ. Για να ανταποκριθούμε ακριβώς σε όλα αυτά τα ζητήματα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όμως και ρωτάω την Κομισιόν εδώ, δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε ε, μια σοβαρή εργασία προγραμματισμού και προς το συμφέρον της αλληλείας, χωρίς να ληφθούν υπόψη δραστηριότητες οι οποίες έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στους ελευθερικούς πόρους και στο περιβάλλον και ε, στον οπιθμένα της ε, θάλασσας. Κύριε Πορμοντέζη, καταλαβαίνω βεβαίως ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται το ότι δεν είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες είναι όμως θεμελιώδους σημασίας. Άρα κινδυνεύουμε να έχουμε ε, έναν προγραμματισμό ο οποίος, πώς να σας το πω, θα είναι περίπου ανώφελος. Εάν βρισκόμαστε σε αλευτική ζώνη και ταυτοχρόνως έχουμε δραστηριότητα εξόριξης ε, ε, κοίτασμάτων ή άμμου ή οτιδήποτε ε, και αν δεν υπάρχει διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων τότε πραγματικά και σας το λέω με πολύ μεγάλη ευγένεια δεν φαίνεται να δείχνουμε μεγάλη σοβαρότητα, δεν είναι πολύ σοβαρό όλο αυτό. είναι γεγονό ότι εγώ διαπιστώνω προβλήματα, δεν προσφέρω λύσει και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά όταν έχουμε ε, όταν έχουμε δραστηριότητες όπως είναι ας πούμε ε, ο τουρισμός, όπως είναι η απομάκρυνση της ε, λάσπης του πυθμένα, δεν είναι δυνατόν να μην τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Το σημαντικό είναι να δούμε που βρίσκονται τα σωστά όρια, έστω και αν την τελική απόφαση, το λέω και το επαναλαμβάνω, θα την ε, ε, πάρουν τα, τα κράτη. Νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να το λύσουμε μαζί το θέμα αυτού του εξαντλητικού καταλόγου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ιζαμπέλ Τωμά, ολοκληρώσαμε την ε, εξέταση των εκθέσεων. Υπενθυμίζω ότι έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις ε, χθε το πρωί στους συντονιστές, οι οποίες ε, έχουν, σας έχουν σταλεί από τη γραμματεία. Βλέπω ότι δεν έχουμε λάβει σχόλια παρατηρήσεις, άρα θεωρούνται εγκεκριμένες οι αποφάσεις αυτές. Να σας υπενθυμίσω ότι η προσεχή εδρία θα λάβει χώρα την 5η Σεπτεμβρίου 2013 από τις 3 μέχρι τις 6.30 εδώ στις Βεξέλλες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Να σας ευχηθώ σε όλους πολύ καλές διακοπές, σε όσους ετοιμάζονται να φύγουν διακοπές και ευχαριστώ πολύ σε όλους. Φαίνεται ότι δεν έχετε καμία διάθεση να φύγετε, μπορείτε να μείνετε αν σας διασκεδάζει το περιβάλλον πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει πρόβλημα.